Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Βεβαίως εγκρίθηκε. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Τράγκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τέταρτο νομισματικό διάλογο του έτους. Όπως θυμάστε, ο προηγούμενος έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα επίσης είχαμε συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Πρόεδρο Ντράγκη και το Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρία πλειοψηφία την έκθεσή του για την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, που διατρανώνει και πάλι την υποστήριξη μας στην νομισματική της πολιτική. Ε, συνάδουν ε, οι ε, ε, δράσει τη με την εντολή της να διατηρεί την σταθερότητα των τιμών, να αποφεύγει ε, πληθωριστικούς κινδύνους και να συνεισφέρει στην οικονομική μεγέθυνση. Ταυτόχρονα εγκρέμε και ένα ψήφισμα που λέει ότι θα πρέπει να αναλυφθούν δράσεις και από άλλους τομείς πολιτικής, να υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική ισορροπία και γενικότερα πιο φιλικές φορολογικές πολιτικές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το τελευταίο νομισματικό διάλογο. Ε, και με το Μάρτιο είχαμε εγκρίνει κάποια μέτρα που εξακολουθούν να υποστηρίζουν ε, και η Κεντρική Τράπεζα μάλλον να υποστηρίζουν δράσεις οικονομικής ανάκαμψης. Ε, είναι μικρά τα βήματα αλλά σταθερά, αργός ο ρυθμός αλλά σταθερός. Στις 20 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο ο πρόεδρος Ντράγκη δήλωσε ότι πρώτοι θα συνεχίσει τα ε, μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης 80 ε, δις και ε, όλα αυτά θα συζητηθούν στο επόμενο Συμβούλιο της Τράπεζας στις 8 Δεκεμβρίου και ενδεχομένω και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική μετά το Μάρτιο βάσει ενημερωμένων στοιχείων και προβολών. Θα παρουσιάσει τη σκοπιά της Τράπεζας όσοι ήθιστε ο Πρόεδρος Δράγκη για τις εξελίξεις οικονομικές και νομισματικές ε, και δύο θέματα που επέλεξαν οι συντονιστές μας, ε, δηλαδή τις επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων στην κερδοφορία των τραπεζών και η λειτουργία του μηχανισμού ε, μη συμβατικών ε, νομισματικών πολιτικών στην Ευρωζώνη. Αυτά τα δύο θέματα ε, θα τα δούμε και σε ακρόαση με ξέχοντες εμπειρογνώμονες. Ο πρόεδρος Δράγκη θα αναφερθεί ιδιαίτερα στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνέπειες του Brexit ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Έχουμε πολλά θέματα λοιπόν. Με μεγάλη περιέργεια θα σας ακούσουμε κύριε Πρόεδρε. Έχετε μέσα στο λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μία εβδομάδα μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τις δραστηριότητες της ΕΚΟΤΟΥ το 2015. Αυτή είναι η τελευταία μου επίσκεψη φέτος, οπότε είναι καλή ευκαιρία να σκεφτούμε ποιες είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις. Το 2016 η οικονομία της Ευρωζώνης ε, ε, απέδειξε ότι είναι ανθεκτική παρά την ανασφάλεια που προέκυψε από την ε, οικονομική και πολιτική σκηνή. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε και στην, η ενίσχυση της Ευρωζώνης αποτέλεσε το βασικό στοιχείο της οικονομικής ανάκαμψης. Στα σχόλιά μου σήμερα θα επικεντρωθώ στις ε, μελλοντικές ε, προκλήσεις ε, σε παγκόσμιο αλλά και σε επίπεδο ευρωζώνης. Και επίσης, τη αιτήση της Επιτροπής σας, θα συζητήσουμε κάποια πράγματα για την βεβαιότητα που προκύπτει από το Brexit και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει από την οπτική της νέας αγοράς. Η παγκόσμια οικονομία, αναμένεται να συνεχίσει την βελτίωσή της, παρόλο που η ανάπτυξη θα παραμείνει αργή, όπως πριν από την, και πιο αργή ίσως από πριν την κρίση. Παρόλο που υπάρχουν ε, στοιχεία ανθεκτικότητας, η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει πολλές σημαντικές ε, και οικονομικές ε, προκλήσεις λόγω της αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα βασικά συμπεράσματα της, του συνάντηση του, της συνάντησης του Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι ότι η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να είναι ο μόνος παράγοντας που θα κινητοποιήσει ισόρροπη ανάπτυξη από μόνη της. Για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, της χρηματοπιστωτικής πολιτικής και της διαφορετικής πολιτικής, χρειάζεται να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και να την κάνουμε πιο συμπεριληπτική. Η ευρωζώνη και η οικονομία της συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, μικρά βήματα, παρά τις ε, αρνητικές επιπτώσεις ε, της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Αυτή η τάση που, που δείχνει να αυξάνεται αναμένεται να συνεχιστεί και κυρίως ε, χάρη στα δικά μας μέτρα πολιτικής. Ιδιαιτέρως η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων μας και οι ε, ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού και οι, πιο, οι δυνατότητες ε, ε, αναχρηματοδότησης των δανείων έχουν βοηθήσει να υπάρξει χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Επίσης, οι βελτιωμένες συνθήκες είναι, βοηθούν όταν κανείς θέλει να λάβει ένα δάνειο από την τράπεζα ή αν θέλει να εκδώσει νέα ομόλογα. Οι μικρές επιχειρήσεις επίσης ε, υποφελούνται και λόγω του χαμηλού κόστους δανεισμού από τις τράπεζες και χάρη στην αυξημένη δυνατότητα των ε, τραπεζών να χορηγούν δάνεια, ενώ οι μεγάλες ε, εταιρείες συνεχώς ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτές οι συνθήκες ε, βοηθούν την επένδυση και τις, και τις και τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Και αυτό βεβαίως φαίνεται και από την ε, αύξηση του ρυθμού δανεισμού των ε, νοικοκυριών αλλά και των εταιριών. Και επίσης, λόγω και των δράσεων που έχουν αναλάβει άλλοι χαράσσοντα την πολιτική, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη μπορούν να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικά η χαμηλή παραγωγικότητα, η ανάπτυξη, τα κάποια προβλήματα που υπάρχουν στον τροπεζικό τομέα, αλλά και η περιορισμένη πρόοδο στι διαφορετικέ αλλαγέ είναι παλιά προβλήματα που πρέπει γρήγορα να αντιμετωπιστούν. Αυτό θα βοηθήσει να κλείσει, να το κενό που υπάρχει πιο γρήγορα και θα αυξήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης που θα βοηθήσει σε, μεγαλύτε, σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Γνωρίζω ότι η προσοχή των φαρασόντων την πολιτική μας έχει αλλάξει μετά από την, τις επιπτώσεις της ε, ε, χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης πρέπει να ολοκληρωθεί η Ένωση, η Νομισματική Ένωση η οποία βρέθηκε πλέον στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Από τότε οι συνθήκες βεβαίως έχουν διαφοροποιηθεί. Σήμερα η Ευρώπη επικεντρώνεται κυρίως στην ασφάλεια και τα, και τα δύο project χρειάζονται ενωμένη Ευρώπη, χρειάζονται συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει καλύτερα να προστατεύσει τον εαυτό της εάν έχει σταθερή και ανθεκτική οικονομία. Και για το λόγο αυτό, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ε, τροτότητες που προκύπτουν από την ατέλεια που την διέπει αυτή τη στιγμή. Ένα επίσης σημαντικό δίδαγμα από την κρίση αυτή είναι ότι ένα μισοχτισμένο σπίτι δεν είναι ποτέ σταθερό. Πάντα κινδυνεύει. Η πρόοδος λοιπόν χρειάζεται σε όλες τις ενώσεις που έχουν καταγραφεί στην ε, έκθεση των ε, πέντε προέδρων. Αυτή η Επιτροπή παίζει έναν ε, πολύ σημαντικό ρόλο στο να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται σημαντική πρόοδο στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο, στου τρέχοντε νομοθετικού φακέλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει επίση ηγετικό ρόλο στα πλαίσια τη προετοινόμενη αναδιατύπωση των νομοθετικών πυλώνων για τα ενιαία λογιστικά βιβλία, ε, για τις κεφαλαιακές, ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσει και επίσης η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσει θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Τώρα, ε, επιτρέψτε μου να στραφώ στις ε, συνέπειες του Brexit, που εσείς μου ζητήσατε να αναφέρω λεπτομερώς. Και για την Ευρωζώνη, αλλά και για, την, ε, για τον Εμένο Βασίλειο, η ενιαία αγορά ήταν ένας πραγματικά θεμελιώδης άσος στο μανίκι της Ένωσης, που συγκερνά τις ευρωπαϊκές οικονομίες Κάτι που μας οδήγησε, βοήθησε συγγνώμη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σημαντικά κέρδη και να καλύψει καλύτερα τη ζήτηση. Για τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η δυνατότητα να ε, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε μια διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή αγορά είναι ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία. Επίσης, η νέα αγορά καθιστά δυνατόν για τις επιχειρήσεις να υποφεληθούν από την συμπληρωματικότητα των διαφόρων ε, τοποθεσιών ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, κομμάτι της αλυσίδας αξιών. Επίσης, η ελεύθερη διακίνηση ατόμων εξασφαλίζει ότι ο καθένας μπορεί να αναζητήσει μια θέση εργασίας εκεί που υπάρχει συγκεντρωμένη οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, τα οικονομικά κλάστερς ε, εποφελούνται από τη δυνατότητα να προσλάβουν ε, πολίτες από όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ενωμένο Βασίλειο έχει εποφεληθεί από, την σημαντική, ε, από τους σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς με την ενιαία αγορά. Μάλιστα, πάνω από 40% των, α, της ε, ε, προσθέμενης αξίας που προκύπτει από τις, ευρω, από τις εξαγωγές προκύπτει από το υπόλοιπο, έρχεται από το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της ενιαίας αγοράς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποτελέσει έναν κόμβο δραστηριοτήτων, τραπεζικών δραστηριοτήτων. Επίσης το ενιαίο διαβατήριο σημαίνει ότι το, οι τράπεζε που βρίσκονται, έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπόλοιπό τη, χωρί να χρειάζεται να έχουν θηγατρικέ εταιρείε στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και βεβαίω το αντίθετο. Αυτό υπονοεί ότι υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση κεφαλαίου και ρευστότητα. Εάν, εάν μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος μιας, πιο, λιγότερο ανοιχτή οικονομίας του ε, Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά και τις άμεσες ξένες επενδύσεις ε, αλλά και άλλους τομείς γινόταν πραγματικότητα θα υπήρχε αρνητική συνέπεια στην καινοτομία και στον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια στην παραγωγικότητα και ίσως ε, στην, στις δυνατότητες κερδοφορίας. Αυτές λοιπόν οι αλλαγέ θα βαρύνουν πρώτα την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και σε ένα μικρότερο βαθμό θα έχουν κάποιες ε, περιορισμένες αρνητικές συνέπειες και στην Ευρωζώνη. Το συνολικό, ο συνολικός αντίκτυπος όμως θα, θα είναι διαφορετικός ανά χώρα, ανάλογα με, τις εμπορικές, με τους εμπορικούς δοσμούς που έχουν με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα η Ευρωζώνη έχει αντιμετωπίσει την, ε, τις αρνητικές συνέπειες του αποτελέσματος του δημοσιοφίσματος ε, με μεγάλη ανθεκτικότητα και χάρη στην προετοιμασία που είχαν κάνει οι κεντρικές τράπεζες αλλά και οι εποπτικές αρχές ένθεν και ένθεν της μάχης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ε, οδήγησε σε μια σημαντική ε, προσπάθεια πρόληψης αποτροπής του κινδύνου, αλλά βεβαίως αυτό δεν κράτησε για πολύ και βεβαίως ε, κατά, τις επόμενες ε, εβδομάδες ε, είδαμε να προκύπτουν διάφορων ειδών εκπλήξεις. Επίσης, ο δείκτης οικονομικών, οικονομικής ικανοποίησης της Ευρωβουλώνης μειώθηκε τον Αύγουστο, αλλά κατα, ανέκτησε τα επίπεδά του τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομική δραστηριότητα επίσης έχει παραμείνει, έχει δείξει ενθεκτικότητα λόγω ακριβώς της άξης της κατανάλωσης. Ταυτόχρονα η ανασφάλεια έχει μειωθεί σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αλλά και, την, και το νόμισμα τη Στερλίνα. Η οικονομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικώ αναμένεται να επιβραδυνθεί. Είναι δύσκολο βέβαια να προβλέψει κανείς την, τις ακριβείς οικονομικές επιπτώσεις της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από τις αποχώρησεις του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα γίνει αυτό, την πρόοδο, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ε, σαφήνεια για την διαδικασία των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ανασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, Θέλω να είμαι σαφή. Ενώ το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της χώρας στην ενιαία αγορά, η ενιαία αγορά δεν μπορεί να πάει πίσω. Είναι σημαντικό η αξιοπιστία της και η ομογένεια των κανόνων της ε, και η εφαρμογή τους να διατηρηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες και για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών που έχουν ενισχυθεί σημαντικά από το 2008. Είναι μάλιστα ουσιώδου σημασία να ενισχύσουμε περαιτέρω και να αναπτύξουμε την ενιαία αγορά. Στον τομέα τώρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Η ενιαία αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υποστηρίζεται πλέον από τον ενιαίο κώδικα κανόνων για τις τράπεζες και τα εποπτικά ιδρύματα. Εντός της Ευρωζώνης έχουμε προχωρήσει και άλλο με την Τραπεζική Ένωση. Βεβαίω δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλο τη διαδικασία. Α πούμε, ε, η οικονομική ολοκλήρωση μέσω μια πλήρου ένωση κεφαλαίου αγορών θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τι ε, χρηματοδοτικέ ε, πηγέ για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε βοηθώντας τον, τον το διαμερισμό κινδύνου για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω εδώ λέγοντας ότι είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ότι κάποιες ε, έρευνες που έγιναν δείχνουν ε, μεγάλη στήριξη για την ε, ενιαία ε, οικονομία παρά τις ε, αντιρρήσεις που υπήρχαν από πολλούς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάντα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Βασικό εκ των οποίων είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτύχει τους στόχους της από την πλευρά των πολιτών της εάν θέλει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να καλύψει βεβαίως το μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας που υπάρχει και οικονομικής μεταξύ των πολιτών. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα λοιπόν χρειάζεται με σημαντικά στέρεα οικονομικά θεμέλια. Για την Ευρωζώνη αυτό σημαίνει ενίσχυση της ε, ε, δυνατότητας ανάκαμψης, ε, οικονομική σταθερότητα και αντιμετώπιση των τροτών σημείων που υπάρχουν ακόμα στην, Ευρωπαϊκή, στην Νομισματική Ένωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως περιμένω τις ερωτήσεις σας. Εγώ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Ντράγκη. Προχωρούμε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Μπάλτς πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας την περασμένη φορά, όταν είχαμε το τελευταίο διάλογο το Σεπτέμβριο, εστίασα στην ερώτησή μου στις συνέπειες του Brexit και ποια ε, είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος. Θα συμφωνήσετε ότι επικρατεί αβεβαιότητα και τώρα αντιμετωπίζουμε και ε, το συνταγματικό δημοψήφισμα στην Ιταλία την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργό Ρέντσι το συνέδεσε στενά το δημοψήφισμα και την έκβασή του με την ίδια του τη μοίρα ως Πρωθυπουργό και επειδή ξέρουμε ότι είναι σε δυσχυμερή θέση, για να το πω έτσι, ήπια το τραπεζικό σύστημα στην Ιταλία, ε, παρακολουθούν τις εξελίξεις όλοι πολύ στενά, όχι μόνο οι πολιτικοί εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και οι οικονομολόγοι και τα χρηματοπιστωτικά. Μπορείτε να τα διαβάσετε στη σημερινή ε, Financial Times. Σας ερωτώ, ανησυχείτε για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που μπορεί να έχει ε, ένα αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία. Ε, μιλώ για τη σταθερότητα ε, του τραπεζικού συστήματος. Ένα άλλο θέμα που κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη πηγή αβεβαιότητας, ακόμα μεγαλύτερη και μεγαλύτερη αδυναμία προβλεψιμότητας. Αυτό αφορά και το διεθνές εμπόριο αλλά και την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη λέγουν ορισμένοι. Εσείς συμμερίζετε σε αυτές τις ανησυχίες και πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη από την εκλογή αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Βλέποντας κανείς τις πρόσφατες εξελίξεις διαπιστώνει ότι ε, για τους επόμενους μήνες θα ε, κυριαρχήσει μια διεθνής αβεβαιότητα και ανησυχία. Μέχρι στιγμής τι βλέπουμε, ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις πάρα πολύ γρήγορα το πρώτο διάστημα, βραχυπρόθεσμα δηλαδή, και από εκεί και πέρα ε, μειώνονται Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αγορές εμφανίστηκαν πιο αθεντικές από ότι θα ανέμενε κανείς πριν από λίγα χρόνια. Και οι ε, χρηματοπιστωτικοί ε, μεσάζοντες ε, και τα ιδρύματα είναι πιο ισχυρά από ότι τα τελευταία χρόνια που παλαιότερα είχαμε και μεγάλες διακοιμάσεις στις τιμές και τις ισοτιμίες. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί μέσω πρόθεσμα, απάντηση είναι όχι. Οι αλλαγές αυτές, όλες, είναι βαθιές, αρκετά. Και πρόκειται να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την πραγματικότητα όχι μόνο των επομένων μηνών, αλλά των επομένων ετών. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε το τελικό αντίκτυπο όλων αυτών. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τι θα πρέπει εμείς να κάνουμε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων αλλού. Με πρώτο και κύριο να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την ανάκαμψή μας, να την ε, εδραιώσουμε, να παγιώσουμε τις βελτιώσεις ε, στην αγορά εργασίας με δημιουργία θέσεων εργασίας Έχουμε εκατομμύρια νέε θέσει εργασία που δημιουργήθηκαν την τελευταία διετία. Να συνεχίσουμε δηλαδή τη δουλειά μα. Δεύτερον, να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση ε, και την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά που είναι τα θεμέλια τα ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, θα πρέπει να διαφυλάξουμε την οικονομική και σταθερότητα. Έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στο μέτωπο αυτό και αυτό που δεν θα θέλαμε τώρα είναι να την καταργήσουμε, να την ξυλώσουμε, να την ε, διαλύσουμε. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ε, τα διδάγματα της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης που είχαμε μια συνεχιζόμενη, διονυζόμενη ε, διατάραξη ε, όλων των κανονισμών που είχαν αποφασιστεί στην αρχή του 2000 και αυτό οδήγησε στη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση και σίγουρα δεν θέλουμε να το δούμε αυτό να επαναλαμβάνεται. Άρα, ισχυρή ανάπτυξη, συνέχιση της εσωτερικής αγοράς, διαφύλαξη της οικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και βελτίωση της αγοράς εργασίας. Να συνεχιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Σας απίθυνα μια γραπτή ερώτηση εγώ για τη συγχώνευση του ε, χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της Γερμανίας. Ε, το London Stock Exchange με την Deutsche Börse δεν έχει άποψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη γραπτή μου ερώτηση. Επανέρχομαι στο θέμα που συζητήσαμε όμως την περασμένη εβδομάδα στην Αλομέλεια και ο συνάδελφος Μπουρκχαρτ Μπάλτς ε, ε, το επανέλαβε. Αυτό είναι ο αντίκτυπος της εκλογής του Ντόναλτ Τραμπ και τι συνέπειες θα έχει στη νομισματική αλλά και την οικονομική μας πολιτική. Την περασμένη εβδομάδα μας είπατε ότι ήταν δύσκολο να προεξοφλήσει κανείς ή να επαληθεύσει απριόρι ε, και τόσο νωρίς. Τι θα σήμαινε αυτό η αύξηση των επιτοκίων, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, όταν είχαμε πάει στην Ουάσιγκτον, ε, στην ετήσια σε τήσεις γενικές συνελεύσεις είδαμε ε, ότι ανησυχούν όλες οι αναδυόμενες χώρες για την ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες αγνοώντας απολύτως τον οικονομικό αντίκτυπο που θα είχε μια τέτοια αύξηση για τις ίδιες τις αναδυόμενες οικονομίες. Κατά κάποιο τρόπο και η Ευρώπη σε αντίστοιχη μοίρα βρίσκεται. Δηλαδή εγώ δεν φρονώ ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας ή η αντίσταση, η αφεκτικότητά της ε, μπορεί να αντισταθεί στη ΦΕΔ αν αρχίσει να ανεβάζει τα επιτόκια. Ερωτώ λοιπόν, εσείς πώς αναλύετε τον αντίκτυπο αυτό στην πραγματική οικονομία και στην νομισματική της Ευρώπης, ενδεχόμενης αύξηση των επιτοκίων δηλαδή στη ΣΥΠΑ. Και δεύτερον, είχατε την ευκαιρία από την εκλογή του κυρίου Τραμπ να συζητήσετε με τον ομόλογό σας, τον κύριο Μπερνάνκη της ΦΕΤ, για το πώς ε, ε, πρόκειται να εξελιχθούν όλα αυτά. Ε, ε, Έχει αλλάξει ε, ο κυβερνήτης της ΦΕΔ. Είναι η κυρία Γιάννη. Ναι, ναι, συγγνώμη, λέει η κυρία Περές. Έχει φύγει ο Μπερνάκη. Έλεγα λοιπόν και για τον νόμο Dodd Frank θα αφισβητηθεί, θα το θέσετε υπόψη της ομολόγου σας από τη ΦΕΔ. Well, um, first let's, let's observe that... Κύριε Ντράγκη. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι η ανάκαμψη στι ΗΠΑ βρίσκεται σε διαφορετική φάση σε σχέση με την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, στι ΗΠΑ η ανάκαμψη έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Κατόπιν τούτο, επειδή διαφέρουν οι συνθήκε, Να δούμε λιγάκι ποια θα είναι η πολιτική της νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια. Να πω όμω ότι αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι μόνο τα επιτόκια, αλλά αυτά που αποκαλούμε οι χρηματοπιστωτικέ συνθήκε, δηλαδή επιτόκια, ε, ισοτιμίες, ε, χρηματιστήρια, ε, αγορέ ομολόγων, κρίση στον τομέα αυτό, όλα αυτά παίζουν ρόλο στη συνάντησή μας για θέματα νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου θα αξιολογήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και που θα επιτρέψουν στο Συμβούλιο να διαφυλάξει σε μεγάλο βαθμό τις νομισματικές εκείνες συνθήκες που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουμε την ε, διακύμανση του ε, πληθωρισμού σε επίπεδα γύρω στο 2% μέσω σταθμικά. Όσον αφορά τη δεύτερη ερωτήσή σας, κοιτάξτε, η απλά όχι. Δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα ε, μέχρι σήμερα να συζητήσω με τον ομόλογό μου από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ με την κυρία, την ομολογώ μου όπως είπαμε προηγουμένως. Ε, σύντομα όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τη στάση που υπάρχει σε σχέση με τους κανονισμούς. Γιατί θα υπάρξουν αρκετές συναντήσεις ε, στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, ε, συναντήσεις κατά τους επόμενους μήνες όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα να δούμε ποια θα είναι η ρυθμιστική ας πούμε στάση της νέας κυβέρνησης. Ο κύριο Μπραντ Λούκε έχει το λόγο. Καλημέρα κύριε Τράγκε. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Και πάλι λοιπόν καλημέρα σας και επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά. Έχετε βάλει τα ακουστικά, είναι εντάξει. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας ε, κάνω μια ερώτηση για το πρόγραμμα Corporate Sector Purchases της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2016. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα αγοράς ε, θα δημοσιεύονται στοιχεία και συγκεκριμένα κάθε εβδομάδα όσον αφορά τα ομόλογα ε, των τραπεζών που συμμετέχουν, των πέντε κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Διαπιστώθηκε τώρα ότι στην ιστοσελίδα αυτών των κεντρικών τραπεζών κάθε εβδομάδα αναφέρονται μεν τα στοιχεία, τα επίκαιρα, όμως τα στοιχεία τα παλαιότερα από προηγούμενες εβδομάδες, αυτά δεν εμφανίζονται πουθενά. Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, η Deutsche Bundesbank, παρότι τη ζητήθηκε, αρνήθηκε σε έναν ερωτώντα να διαθέσει στοιχεία παλαιότερων προθεσμιών παλαιότερων εβδομάδων. Εγώ λοιπόν ως ε, Ευρωβουλευτής ε, προσπάθησα να αποκτήσω αυτά τα ιστορικά αν θέλετε στοιχεία και θέλησα επίσης να πω ότι και οι υπόλοιπε πέντε κεντρικές τράπεζες και αυτές το έκαναν. Ε, δυστυχώς όμως η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, η Bundesbank δεν έχει δώσει αυτά τα στοιχεία. Και σας ερωτώ, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί η Bundesbank στοιχεία τα οποία είχε δημοσιεύσει μετά όμως τα απέσει από την ιστοσελίδα της, γιατί δεν τα διαθέτει αυτά σε ενδιαφερόμενους. Και μήπως και εσείς πιστεύετε ότι όσον αφορά τις κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στην ΕΚΤ, δεν θα πρέπει για όλες να ισχύει η ίδια διαφάνεια. Άρα δηλαδή θέματα που ενδεχομένω αφορούν τις τράπεζες και ενδιαφέρονται σε σχέση με την Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, να μπορούν οι άλλες κεντρικές τράπεζες να τα αποκτήσουν. Κύριος Ντράγκη, επιτρέψτε μου να πω κάτι σχετικά με το πρόγραμμα αυτό το Corporate Bond. Ε, κοιτάξτε, έχουμε τις ε, εταιρείε που διαπιστώνεται ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όπως κατά τα μέσα του ε, 11, αλλά υπάρχει και μία σημαντική αύξηση. Τώρα πλέον ε, όπως σας είπα υπάρχει αυτό το επίπεδο. Κοιτάξτε, αυτό που με ρωτήσετε δεν το ξέρω καλά. Θα το ψάξω και αν δεν σας πειράζει να σας απαντήσω σε γραπτή μορφή. Για να είμαι σίγουρος ότι θα τα ψάξω σωστά. Κοιτάξτε, επιτρέπτε μου να σας ερωτήσω. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω συμπληρωματικά. Όσον αφορά το θέμα της αρχής, επέστε μου τουλάχιστον για το θέμα της αρχής, δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι όλες οι συμμετέχουσες κεντρικής τράπεζες θα πρέπει όλες να διασφαλίζουν έναντι του πολίτη το ίδιο επίπεδο διαφάνειας. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει και η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα να δημοσιεύει και αυτή η στοιχεία που δημοσιεύουν άλλες κεντρικές τράπεζες χωρίς καν να το κάνουμε θέμα. Κύριε Δράγκη, συμφωνώ σε επίπεδο αρχή, αλλά δεν καταλαβαίνω, μάλλον δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε αυτό η Deutsche Bundesbank. Και επιτρέψτε μου να σα δώσω σε γραπτή μορφή, όπω σα είπα, μία απάντηση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο κύριο Πέντ Λούκε. Ευχαριστώ, κύριε Σιλβέ Γκουλάρ. Καλημέρα, Πρόεδρε, στα Ιταλικά και στα Γαλλικά. Θα μιλήσω γαλλικά. Το Brexit, όπως και η εκλογή του Donald Trump στι Ηνωμένε Πολιτείες, καθώς και όλα τα θέματα ε, που έχουν μείνει εκκρεμοί για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης μου φαίνεται ότι αναδεικνύουν το ίδιο θέμα που είναι η συλλογική κυριαρχία της Ευρωζώνης. Συλλογική ε, μιας ε, ζώνης που έχει το ίδιο νόμισμα. Και στο βαθμό που ελέγχουμε εμείς τα εργαλεία που μπορούν να διακυβεύσουν τη σταθερότητά μας ε, η κερδοφορία των τραπεζών, ε, η ύπαρξη μια αυτόνομη τραπεζική ε, οντότητα στην Ευρωζώνη απακιστρωμενη από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασχολείται με αυτό το θέμα και θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να έχουμε πιο βαθύ διάλογο, δηλαδή μια στρατηγική θεώρηση και σκέψη. Συχνά με την ΕΚΤ συζητούμε θέματα τεχνικά και το εκτιμούμε βαθύτατα γιατί μα διαφωτίζει, αλλά να έχουμε πιο στρατηγική θεώρηση αυτή τη νομισματική κυριαρχία. Και κάποια στιγμή μήπω θα ήταν σκόπιμο να ε, επιστήσουμε την προσοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που από τη φύση του είναι αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων των χωρών και στερούνται τη συλλογική σκέψη αυτή, δυσκολεύονται να δουν αυτό συλλογικά. Ακριβώς όπως το θέσατε, επειδή υπάρχουν πολλές αναταραχές τώρα και αναταράξεις παγκοσμίω, μήπως θα μπορούσαμε να δούμε πιο πολύ και πιο στρατηγικά αυτό το θέμα από κοινού. Ευχαριστώ. Τους επόμενους μήνες και στις ε, επερχόμενες διαπραγματεύσεις ε, ε, μετά από το Βρετανικό δημοψήφισμα θα τεθούν ζητήματα σίγουρα κυριαρχίας στις υποδομές, στις πληρωμές μας, στο σύστημα clearing κτλ. Άρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο και όλα αυτά τα θέματα. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές το εξής. Έχουμε μια πολιτική για ένα σύστημα ε, πληρωμών, αλλά όχι για τις υποδοπές μέσα των αγορών. Αυτό δεν έχει να κάνει ε, με το Brexit, αλλά έχουμε την οδηγία EMIR ε, και αν κάποιο πρέπει να το αλλάξει αυτό ή θέλει να το αλλάξει, να σε εσά, του νομοθέτε. Είτε θα αλλάξετε το, καταστατικό τη ΕΚΤ, είτε την νομοθεσία και την οδηγία αυτή. Έχετε δίκιο όμω ότι θα υπάρξουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Εάν επιθυμούμε σταδιακά να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Είναι πολύ ευάλωτη σε πολλά σημεία η νομισματική ένωση και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Σε ποιο βαθμό μπορούν οι χώρες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών συγκεντρώνοντας, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους και τους πόρους τους και με συγκυριαρχία στους τομείς που θεωρούν εκείνα ε, τα κράτη ε, απαραίτητους. Ή συνεχίζει κάθε χώρα τη δική της πορεία η απάντηση είναι ότι όσο πιο υπερεθνικό είναι το πρόβλημα, τόσο πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό θα είναι να απαντηθεί από κοινού. Αυτή είναι μια προοπτική ρεαλιστική, πραγματιστική που είχαν και οι πατέρες ιδρυτές της ευρωπαϊκής κοινότητας όταν την ίδρυσαν. Ευχαριστώ. Thank you, Ματίας. Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, μιλούμε πολύ για το Brexit και τους, ε, τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Και ήθελα να σας ε, θέσω ευθέως ένα ερώτημα σήμερα. δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Brexit μόνο αποκομμένο από όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να δούμε και τα δικά μας εσωτερικά θέματα. Έχουμε δει τους τελευταίους μήνες πάρα, πολλά, πάρα πολλούς, πάρα πολλούς στοχασμούς για το κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό χαλάρωσε, θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες είναι μία από τις α, λίγες πολιτικές της Ευρωπαϊκής που ενισχύουν την οικονομία. Αλλά ξέρουμε ότι ε, αυτά τα ωφέλιμα αποτελέσματα ε, δυστυχώς ε, έμειναν στη δεύτερη μοίρα λόγω των ε, πολιτικών λιτότητας. Οι αγορές ομολόγων στις τράπεζες έχουν επιτρέψει σε χώρες όπως η Πορτογαλία να βοηθούν σε ό,τι αφορά το χρέος, αλλά η ΕΚΟΤΟΥ στέλνει συνεχώς το μήνυμα ότι θέλει να εγγυηθεί τη σταθερότητα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν δεν λέει κανείς τι, τι πρόκειται να κάνει, δημιουργεί περισσότερη αστάθεια στις αγορές και ανασφάλεια. Και ε, στο τέλος ε, γίνεται προσπάθεια να αποφευθούν ας πούμε, τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Η δική σας δράση ποια θα είναι ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε παλαιότερες περιστάσεις είχατε πει ότι το πρόγραμμα θα συνεχίσει και γι' αυτό θα χρειαστεί ωστόσο οικονομική ανάπτυξη. Αλλά ούτε το πρόγραμμα βλέπουμε να συνεχίζεται, ούτε οικονομική ανάπτυξη έχουμε. Οπότε αναρωτιέμαι, γιατί δεν έχετε ήδη ανακοινώσει την συνέχεια του α, προγράμματος αυτού α, αποστηγής χαλάρωσης μέχρι, μετά το Μάρτιο. Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από, εσάς, από εμένα πώς επιδρά η αβεβαιότητα. Ευχαριστώ. Ναι, να πω και πάλι, απαντώντας την ερώτησή σας. Αυτό που είπα στην αρχή. Στην ε, συνεδρίαση για την νομισματική πολιτική το Δεκέμβριο θα αξιολογήσουμε τις διάφορες επιλογές που θα επιτρέψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διατηρήσει την ε, δυνατότητα, τον ε, βαθμό παρέμβασης που μπορεί να έχει έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τη σύγκληση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό για να παραμείνουν σε επίπεδα κοντά στο 2% σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα έχουμε λίγη ακόμη ανασφάλεια, βεβαιότητα. No? I think uh, I, I've said that. Okay. Please, you have time. Αν έχετε χρόνο, αν θέλετε. Ω, όχι, Πρόεδρε. Δεν, ε, δεν θέλω να το συνεχίσουμε, αλλά ε, ε προ, αναφέρατε δύο προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις θα οδηγήσουν στην αναστολή του προγράμματος, αλλά καμία από τις δύο δεν πληρείται προς το παρόν. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε σαφώς. Αυτό ακριβώς η ασάφεια είναι που δημιουργεί την αστάθεια στην Ευρωζώνη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί ε, επιλέγετε να την συνεχίζετε. Όχι, δεν έχουμε την ίδια οπτική των πραγμάτων. Αυτή είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ληφθεί το Δεκέμβριο οι όροι κάτω από τους οποίους θα ληφθεί η απόφαση, αν ακούσατε αυτά που είπα, είναι αυτοί ακριβώς που σας ανέφερα. Μπορώ να τα ξαναπώ αν επιθυμείτε. Στην συνάντηση λοιπόν της νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου θα αξιολογήσουμε τις διάφορες επιλογές που θα επιτρέψουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαφυλάξει τον ουσιώδη βαθμό ε, νομισματικής ε, διευκόλυνσης που είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει τη μόνιμη ε, προσέγγιση των δικτών του πληθωρισμού που θα τους διατηρήσει σε ένα 2% σε ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μου απαντήσατε με ένα πολύ γραφειοκρατικό τρόπο σε ένα διοικητικό ερώτημα, αλλά εντάξει. We will see very soon. Um, λοιπόν, θα δούμε πολύ σύντομα. Μόλις Σκοτ Κότο. Πρέπει να πω ότι είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και ήμουν κατά της ένταξης της Βρετανία στο ευρώ για πολιτικούς ε, λόγους γιατί θεωρούσα ότι δεν υπήρχε ε, πολιτική υποστήριξη και συμφωνία μεταξύ των κρατών μερών να υποστηριχθεί ένα ισχυρό νόμισμα. Η κατάσταση όμως με το Brexit με έκανε να αναθεωρήσω και επειδή ξέρετε εγώ ήμουν πάντα οπαδός της Τερλίνας, ε, χρειάστηκε να κλονιστώ όταν το ξανασκέφτηκα. Η απόφαση να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εσωτερική αγορά πιστεύω ότι ε, υπονόμευσε τη διεθνή αξιοπιστία της Τερλίνας. Και επίσης ε, δεν είναι πλέον και ένα νόμισμα στο οποίο καταφεύγει κανείς για αποθεματικά. Ε, τελικά, εάν φύγει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει. Εγώ παραμένω στη θεώρησή μου ότι δεν υπάρχει αρκετή πολιτική στήριξη και θα είναι ε, ασταθέ και ασθενέ και το ευρώ ω νόμισμα. Αλλά από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Μπορεί να μου πείτε ότι δεν είναι πολιτικά αυτά τα θέματα, αλλά είναι. Υπάρχουν απειλέ για ε, τι θέσει εργασία στο ΣΥΤΙ, ε, αν σταματήσει να συμμετέχει στο σύστημα πληρωμών και διακανονισμών ε, η Βρετανία. Για να πετύχει το ευρώ χρειάζεται πολιτική στήριξη αλλά και στήριξη από τους πολίτες και την κοινή γνώμη. Εσείς πώς το βλέπετε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί, πώς να επιχειρηματολογήσουμε, ιδιαίτερα και εν ώψη της ε, ακροδεξιάς που σηκώνει κεφάλι και απειλεί όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ως νέο νόμισμα. Εσείς πώς βλέπετε τον αντίκτυπο του Brexit για την Στερλίνα. Συμφωνείτε με τη Σταρεμπούρς ότι θα πρέπει να παραμείνει ένα παγκόσμιο νόμισμα για αποθεματικά. Θα παραμείνουν θέσεις εργασίας στη ΣΥΤΗ και τι θα σημαίνει αυτό για άλλο το χρηματοπιστωτικό τομέα στην Βρετανία. Συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, πολλά πράγματα με ρωτάτε και πολύ ενδιαφέροντα αλλά πολύ δύσκολα. Και όπως είπατε, ίσως εγώ να μην είμαι ε, ο κατάλληλος για να τις απαντήσω, γιατί αυτά που με ρωτάτε ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητές μου. Σε πολλές από τις ερωτήσεις που κάνατε η απάντηση είναι μία. δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Δεν το γνωρίζουμε απλούστατα. Για ποιο λόγο. Διότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς με ποιον τρόπο θα οριστικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις, ποια θα είναι η τελική τους μορφή και πόσο θα κρατήσουν έτσι χρονικά. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι όσο περισσότερο τραβήξουν σε μάκρος ε, και διονίζονται, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και βεβαιότητα και ανασφάλεια. Να κάνω ένα βήμα πίσω. Για τη σημερινή κατάσταση, πριν από λίγα χρόνια, τι συνέβαινε. Το City του Λονδίνου καταλάβαινε και έκανε ε, ποιες είναι οι μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και στον υπόλοιπο κόσμο αντίστοιχο όγκο συναλλαγών είχε μόνο η Νέα Υόρκη. Αυτό πώς θα αλλάξει τώρα. Δεν το γνωρίζουμε. Θα ε, ξαναδημιουργηθεί κάπου αλλού αυτό, ούτε αυτό το γνωρίζουμε. τα κέρδη που είχαμε από τις οικονομίες κλίμακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι θα γίνουν, θα επαναληφθούν αλλού ή μήπως θα μετακινηθούν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Όλα αυτά τα ζητήματα τα κοιτάμε, αλλά επίσης κοιτάμε και να μας πει τι θέλει η Βρετανική κυβέρνηση. Να μοιραστεί τα σχέδια και τις προθέσεις της, όχι μαζί μας, με τους πολίτες τους και να δούμε τι θα πούνε εκείνοι πριν αποφανθούμε εμείς να πούμε ποιες είναι δικές μας απόψεις από αυτόν. Ε, Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρόσφατα εκτός από το δημοψήφισμα αυτό για την Ιταλία, για το οποίο συζητάμε, ε, θα υπάρξει ε, την ίδια μέρα, θα υπάρξουν και εκλογές ε, στην Αυστρία. Και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν δηλώσεις ε, από τον υποψήφιο του Παρτίντο Λιμπερτά. Σύμφωνα με ε, δημοσκοπήσεις έχει περίπου το 50% και με βάση αυτές τις δηλώσεις αν η Ευρώπη συνεχίσει με μια συγκεντρωτική πορεία η Αυστρία με εκείνον ε, πρόεδρο πλέον θα είναι αναγκασμένη να διοργανώσει δημοψήφισμα για την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα είπε κάποιος ο οποίος λέω Βεβαίω στι δημοσκοπήσει σκυγεντρώνει πάνω από 50%. Άρα δηλαδή υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να κυβερνήσει την Αυστρία. Και ρωτώ, η κεντρική, η εκτε προετοιμάζεται για τέτοιου είδου σενάρια στην Αυστρία. Ε, δηλαδή να αποφασίσει η Αυστρία αν θέλετε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά κάποιον τρόπο να σπάσει τη ραχοκοκαλιά της Ευρωζώνης. Και άλλη μία πολύ γρήγορη ερώτηση ε, σχετικά με τις τράπεζες στην Ιταλία, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίματος, είναι κάπως ευαίσθητη η κατάσταση. Και θέλω να μου πείτε, στην περίπτωση κατά την οποία ε, προκύψουν ε, δυσκολίες κεφαλαιακές όσον αφορά στις τράπεζες, θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί κάποιο σύστημα που να υπάρχει στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της κρίσης. Η ΕΚΤ έχει σκεφτεί να εφαρμόσει κάποια λύση έτσι ώστε να αποφύγει να υπάρξει ε, κάποια κρίση η οποία θα μπορούσε να αποβεί και συστημική. Επιτρέψτε μου να πω, όσον αφορά στην πρώτη σας ερώτηση, να πω το εξή. Το εξή, ότι χωρίς να θέλω να εστιάσω την προσοχή μου σε μία και μόνο χώρα, εμείς βλέπουμε ε, τα ευρωσκεπτιστικά κόμματα τους, ε, τα τελευταία χρόνια έχουν αέρα στα πανιά τους και από ό,τι φαίνεται οι πολίτες ε, δεν ανθίστανται κατ' ουσίαν στο να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε, στην, στην, στην Ευρώπη. Εκείνοι όμως λένε κάτι διαφορετικό. Λένε ότι θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στοχεύσει στις βασικές τους ανησυχίες, να τους προστατεύσει από οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ασφάλειας και να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που να έχουν μια σαφή διεθνή διάσταση, όπως είναι η μετανάσταυση, θέματα ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, τρομοκρατίας, τέτοιου είδους θέματα. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, αν θέλετε, οι πολίτες στηρίζουν το ενιαίο νόμισμα ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς. Η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Βέβαια, η υποστήριξη για τους εθνικούς φορείς, πράγματι αυτή έχει αμβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Άρα φαίνεται ότι οι πολίτες ε, χαρακτηρίζονται από μια έντονη επιθυμία να υπάρχουν λιγότεροι συστημικοί κινδύνοι στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα στην ΕΚΤ, οι αλλαγές αυτές οι οποίες λαμβάνουν, από, λαμβάνουν χώρα στις απόψεις των πολιτών. Θα δούμε βέβαια τώρα τι θα γίνει, αν αυτές θα είναι μακροχρόνιες απόψεις ή βραχυπρόθεσμες. Εγώ πιστεύω το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε πολιτικές που ενισχύουν την ανάκαμψη, βελτιώνουν τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και διαφυλάσσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και έτσι απαντώ στη δεύτερη ερώτησή σας για τις Ιταλικές τράπεζες. Δηλαδή η ΕΚΤ δεν έχει προβλέψει ειδικού κανόνες, αλλά ούτε είναι και δική μας αρμοδιότητα το να παρέμβουμε. Υπάρχουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν οι οδηγίες και η καλύτερη συνεισφορά που θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΚΤ είναι η εποπτεία ως προς το ότι οι κανονισμοί και είναι σωστά σχεδιασμένοι και εφαρμόζονται με σαφήνεια. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μπερνάρ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ντράγκη. Καλημέρα σας. Δύο βασικά ζητήματα. Το ε, πρόγραμμα αυτό που, ασκείτε, που υιοθετείτε ε, είναι ε, για την ενίσχυση της οικονομίας από το 2012. Έχει έρθει η ώρα του απολογισμού. Πέρα από τα δώρα που κάνει στις τράπεζες η ΕΚΤ, στόχο σας είναι να αυξηθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επιτευχθεί, έχετε γενικέ στρατηγικέ να μα δώσετε στατιστικέ και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το δεύτερο ε, αφορά τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας και τη διαχείρισή του. Ε, Πρόσφατα αμφισβητήθηκε η λειτουργία του. Τι φρονείται για την έκθεση αυτή. Φαίνεται ότι δεν έχει τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπίσει τις νέες υποχρεώσεις εποπτείας και καμιά φορά είναι κακή οργάνωση ή υπερβολικός ο φόρτος εργασίας για το προσωπικό. Και επαφίεται πολλές φορές στις εθνικές αρχές για να κάνει ε, αυτός ο πυλώνας ε, το έργο του. Ο δεύτερος πυλώνας ε, δεν εφαρμόζεται όπως φαίνεται από την Ιταλία και τη Γερμανία και ο τρίτος πυλώνας δεν πρόκειται ποτέ να ε, υλοποιηθεί γιατί δεν το θέλει η Γερμανία. Ε, άρα το SSM έχει αποτύχει εκτρά γιατί δεν δίνεται στις χώρες την κυριαρχία τους για τη διαχείριση των εθνικών τους τραπεζικών συστημάτων. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω την απάντησή σας. Η πρώτη απάντηση είναι ότι τα προγράμματα Τέλτρο και των εταιρικών ομολογών έχουν επιτύχει σε μεγάλο βαθμό ε, το στόχο τους για την πραγματική οικονομία. Το είπα και προηγουμένως, αυξάνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη και τώρα έχουμε επανέλθει σε επίπεδο του 2011. Βλέπουμε και το πρόγραμμα για τα εταιρικά ομόλογα έχει απελευθερώσει και χώρο και συχνά μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Μήπως η πολιτική μας είναι υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Όχι. Ε, το πρόγραμμα Corporate Bond έχει ε, ε, δώσει περιθώριο και ανάσα στις τράπεζες, στους ισολογισμούς τους για να δανείζουν περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το βλέπουμε από στοιχεία μήνα με το μήνα. Για το άλλο θέμα που ρωτήσατε για την έκθεση ε, του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρεστε σε αυτή. Να σας πω ότι εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και πράγματι μας βοηθά για να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις ανησυχίες που όντως έχουν εκφραστεί σε αυτή την έκθεση. Δίνει μια νέα προοπτική ουσιαστικά και εντοπίζει ε, το μυς που χωράνε βελτιώσεις. Τούτον όμως λεχθέντων δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο SSM είναι καταπληκτικό επίτευγμα. Το να στήσει ένα σύστημα ενιαίο ε, εποπτείας για 19 χώρες και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τράπεζες μέσα σε μία διετία ε, δεν είναι και ευκαταφρόνητο. Βέβαια δεν είμαι εγώ αντικειμενικός παρατηρητής, ε, άρα τα λόγια μου έχουν την αξία αυτή που έχουν. Συμφωνούμε με το ελεγκτικό συνέδριο στις εκτιμήσεις τους για την ανάγκη να στελεχωθεί καλύτερα ο SSM. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερους πόρους και θα γίνει και μια συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, της ΕΚΤ πάρα πολύ σύντομα πριν ε, το τέλος του έτους ακριβώς για αυτό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα λέγει το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θέτει το ζήτημα που αναφέρατε, στο, υπενυχτήκατε, ότι επί τόπου ε, επιθεωρήσεις και αλλαγή γίνονται κυρίως από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Μα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν πρέπει κάποιος να προσλαμβάνει χιλιάδες επί χιλιάδων ε, σε μικρό διάστημα, ε, υπάρχει και κίνδυνος για λάθη. Τώρα έχουν προσληφθεί πάνω από χίλιοι υπάλληλοι. Δηλαδή ε, κάπως υπάρχει ένας καταμερισμός και ε, ανατίθεται και έλεγχη στις εθνικές αρχές. Ο SSM όμω δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόνη της. είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Μπορούμε βέβαια να αυξήσουμε σταδιακά τις επιθεωρήσεις ε, που κάνουν επιτόπου οι δική μας ε, και της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά δεν είναι ε, μια μεγάλη πίτα στη Φραγκφούρτη που τα αναλαμβάνει όλα αυτά. Έχουν και γνώση και πείρα και ιστορία οι εθνικές αρχές και το αξιοποιούμε. Επίσης, κάτι άλλο που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε είναι ότι πολλές φορές είναι κοινέ οι ομάδες των επιθεωρητών, ακόμα και αν υπό την αιγίδα και επικεφαλής είναι κάποιοι εθνικοί ελεκτές. Και πολύ συχνά υπάρχουν και διάφορες εθνικότητες, δηλαδή επιθεωρητές από τη Γερμανία που ελέγχουν τις τράπεζες σε άλλες χώρες, όπως ε, και από την Ιταλία και τη Γαλλία. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πρέπει να έρθει κάποιος από τη Φραγκφούρτη για να εγγυηθεί ότι είναι ανεξάρτητος ο έλεγχος και αμερόληπτος. Εν πάση περιπτώσει. Δεν βοηθάει το σχόλιο αυτό. Μάλλον μας βοηθάει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για να αυξήσουμε το προσωπικό. Ε, λένε και άλλα ε, στην έκθεσή τους, αλλά δεν αναφερθήκατε σε αυτά του ελεκτικού συνεδρίου, οπότε δεν θα απαντήσω. Αν με ρωτήσει κάποιος, έχω να πω κι άλλα. Thank you. Danuta Hubner. Η Ντανούτα Χόμπνερ, ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα έχω. Ένα για την ε, ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, γιατί μπορεί να υπάρχουν ίσως κάποια πρώτα αποτελέσματα ή ίσως κάποια νομοθεσία και ίσως ε, μπορούμε να έχουμε την αρχή της διαδικασίας έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε κάποιες αλλαγές για την ε, χρηματοδότηση της οικονομίας. Δεν ξέρω βέβαια ότι θα έχουμε απομάκρυνση από την ε, χρηματοδότηση με βάση τις τράπεζες τόσο γρήγορα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Μπορούμε βέβαια αυτό να το δούμε και από την μακροπροληπτική οπτική, μπορούμε να το δούμε και από την οπτική του αντικτύπου στην αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα της νομισματικής πολιτικής. Δεν ξέρω αν το έχετε ήδη σκεφτεί κατά αυτόν τον τρόπο, ε, τι θα σημαίνει δηλαδή ε, για την νομισματική πολιτική η Ένωση Κεφαλαιογορών. Και επίση, δεύτερη ερώτησή μου. Από καιρού καιρών βλέπουμε στα μέσα μαζική ενημέρωση ε, ότι η ECB μπορεί να μην έχει πια ομόλογα να αγοράσει. αυτό το μείον 0,4 το επίπεδο απόδοσης είναι κάτι που το έχετε επιβάλει εσείς στον εαυτό σα. ουσιαστικά. Οπότε θα μπορούσατε ίσω και να το τροποποιήσετε. Αλλά μήπως μπορείτε να δώσετε λίγη περισσότερη σαφήνεια σε όλη αυτή τη διαδικασία για το πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για το πρώτο σας ερώτημα. Μία από τις εμπειρίες που είχαμε από την ε, οικονομική κρίση είναι ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουμε περισ... διαφορετικές διάβλους ε, μεταφορά της νομισματική πολιτικής στην πραγματική οικονομία και να μην ε, βασιζόμαστε μόνο στην, ε, στο, στο διάβλο των τραπεζών που χρειάστηκε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης γιατί αυτό σήμαινε πάνω από 80% της ε, ε, παρέμβασης. Τώρα έχει, της διαμεσολάβησης, τώρα έχει μειωθεί λίγο. Βεβαίως υπάρχει και δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι κεφαλαιογορές από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Βεβαίως, Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας ε, και ίσως να το ξαναδούμε στα πλαίσια της ακρόασης. Αλλά όπως προχωρούμε από, την, ε, από το τραπεζικό σύστημα στις κεφαλογορές, περνούμε από το τραπεζικό στο μη τραπεζικό ή σκιώδη τραπεζικό τομέα. Και όπως γίνεται αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο ποιος είναι ο κανονισμός της ε, πρόληψης, ποιο είναι το πλαίσιο για αυτόν τον τομέα. Αλλά Αυτό δεν αφορά άμεσα την ε, ε, διαβίβαση της νομισματική πολιτικής, αλλά όντως συμφωνώ ότι βεβαίω θα πρέπει να είναι σωστά λειτουργούσα η κεφαλόγορα, εφόσον βεβαίω δεν υπάρχει κατακρεματισμό. Και γι' αυτό, γι αυτό το σημείο ακριβώς χρειάζονται βήματα τους επόμενου μήνε, τα επόμενα χρόνια, για να δημιουργήσουμε μία κεφαλόγορα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακρεματισμό που εξακολουθεί να υφίσταται. Για το δεύτερο ερώτημά σα, για την ε, ανυπαρξία ε, η σπανιότητα των ομολόγων. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε, αλλά το πρόγραμμα μας είναι αρκετά ευέλικτο, οπότε μπορεί να αναθεωρηθεί, να ξαναχρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε, όπως είπα και πιο πριν, ε, την ε, δυνατότητα, το βαθμό νομισματικής διευκόλυνσης για να επιτύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, επιμένει και καλεί την πολιτική τάξη να δημιουργήσει ε, πολιτικές σε, ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Είπατε ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι ε, το, ο, μόνο, ο μόνος μοχλός που θα οδηγήσει την ανάπτυξη και ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομικές πολιτικές, διαρθρωτικές πολιτικές έτσι ώστε να ενισχύσουμε το δυναμικό της ανάπτυξης. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ υπάρχει κάτι καινούριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πολύ πρόσφατα μία δημοσιονομική πολιτική για τα επόμενα έτη που είναι, που είναι λίγο, έχει ένα, μια, ένα χαρακτήρα διεύρυνσης. Αυτό θεωρείται ότι είναι θετική εξέλιξη ε, αντιστοιχεί στις κλήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. για το 0,5% του ΑΕΠ. Ε, είναι αρκετό αυτό να ενισχύσει, να βοηθήσει την ανάπτυξη. Και επιπλέον, σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο προπολογισμό που έχει εγκριθεί για, τον επόμενο, για το επόμενο έτος δεν δημιουργεί κάποια τέτοια α, επεκτατική πολιτική, αλλά εξακολουθεί να επιμένει στην, στον περιοριστικό δανεισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να πάνε επέκεινα των δημοσιονομικών πολιτικών τους. Και η ερώτηση μου προς εσάς είναι, είναι επιθυμητό για τα κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο δημοσιονομικό στη διάθεσή τους είναι σωστό ή θα μπορούσαν να ε, καλύψουν ή να απαντήσουν σε, αυτό το, σε αυτή την έκκληση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, Βεβαίω σημειώνουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την, ε, ε, για μια πιο σταθερή δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Έχουμε πει και μας το υπενθυμίσατε κι εσείς ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρως, πλήρη την απόδοση των δημοσιονομικών μέτρων πρέπει να συμβάλλουν και άλλα μέτρα και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δημοσιονομικέ πολιτικές ε, θα πρέπει να ενισχύσουν φυσικά, να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ανάκαμψη, αλλά θα πρέπει να είναι συμμορφούμενε με τους δημοσιονομικού κανόνες τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, έμφαση που δίνει στις ε, δημοσιονομικέ αυτές πολιτικές. Έχουμε πει ότι οι χώρε θα πρέπει να επιτύχουν, να έχουν μια πιο φιλική προ το χρήστη δημοσιονομική πολιτική και αυτό αναφέρεται στην ε, ανακοίνωση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει ότι αν μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά την δημοσιονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για τις μελλοντικέ συζητήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει νομικές δεσμεύσεις για τα κράτη-μέλη τα οποία εξακολουθούν να δεσμεύονται από το ε, Σύμφωνο ε, Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Τα σχέδια προπολογισμού για το 2017 των κρατών μελών δείχνουν ότι υπάρχει μια ουδέτερη κατάσταση δημοσιονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση που σημαίνει ισορροπία μεταξύ τη ε, σταθερότητα, τη προβλεπόμενη σταθερότητα και των αναγκών που υπάρχουν. Όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμβολή του κάθε κράτους μέλους ε, ε, τονίζεται στη, στα, που τονίζεται στο, στα σχέδια προπολογισμών ε, δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν που βρίσκονται στο επίπεδο τη μη συμμόρφωση θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να συμμορφωθούν με του δημοσιονομικού κανόνες. Άλλοι πάλι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή του. Οπότε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει το αίτημα της, ε, την έγκριση της Κομισιόν για την ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Ταμείων για τις στρατηγικές επενδύσεις, ε, επέκταση δηλαδή του σχεδίου Γιούκας και βεβαίως προβλέπει στην Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση ε, της Νομισματικής Ένωσης που προβλέπεται για τον Μάρτιο του 2017. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάρκους Φέμπα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω και εγώ δύο σύντομες ερωτήσεις. Αυτή η μία ερώτηση είναι ε, πώς αντιμετωπίζετε τις, ε, τα δάνεια που ενδέχεται να εξελιχθούν σε κόκκινα δάνεια. Γιατί έχει διαπιστωθεί ότι ο τομέας των τραπεζών υποφέρει από αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Άρα δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχει καν αγορά για τέτοιου είδους μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μήπω μπορείτε να μα εξηγήσετε που οφείλεται αυτό και τι μπορεί να γίνει σε ρυθμιστικό επίπεδο και γιατί μόλις το Σεπτέμβρη του 2016 ξεκινήσατε τη διαδικασία διαδικασία των διαβουλεύσεων τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Ε, δεύτερη ερώτηση. Είδα την ιστοσελίδα σα το γράφημα και διαπιστώνουμε εκεί ότι υπάρχει περίπου το επίπεδο του 2012. Εκεί έχουμε φτάσει. Ε, εσείς ανησυχείτε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ιταλία και ακολουθεί μετά και η Ισπανία θεωρούν ότι αυτά τα επιτόκια οι αυτές οι μερίσεις δεκιμάνσεις ε, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Thank you. Uh, on, on MPL, I, I would agree. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα MPL, συμφωνώ μαζί σας. Ε, καταρχήν, αυτό είναι ένα θέμα ε, σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPL όπως είπαμε, ότι είναι ένα θέμα που πρέπει πράγματι να αντιμετωπιστεί σοβαρά, γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί, τον διζημιώνει την κερδοφορία των τραπεζών και τη δυνατότητα των τραπεζών να προσφέρουν δάνεια στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αλλαγές ε, οι οποίες πρέπει να εισαχθούν έτσι ώστε να υπάρχει μια αγορά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπου δεν υπάρχει αυτή. και αυτό απαιτεί να υπάρχουν νομοθετικές αλλαγές για να δούμε πώς είναι δυνατόν να συστήσουμε μια αγορά ε, με τις καλύτερες τιμές για αγορά και πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα περίπτωμα out of court settlements και η συμμετοχή των μεσαζόντων που ε, μπορούν να χειριστούν τα θέματα. Αυτό αλλάζει στα θέματα και σε επίπεδο δικαστηρίων. Σε γενικές γραμμές όμως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι θέμα παρακαταθήκης. Και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, νομοθετικές αλλαγές, αυτές τι κάνουν. Αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Άρα δηλαδή ε, η χρησιμότητα είναι περιορισμένη που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Όσον αφορά την ισορροπία των target του, εκεί έχει υπάρξει βελτίωση και αυτό από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμά μας αγοράς ομολόγων. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που το εξηγούν αυτό. Κοιτάξτε, περίπου το 80% των ομολόγων που αγοράζουν οι κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 80% πωλείται από ε, ιδιοκτήτες που δεν βρίσκονται, δεν ε, εγκαταβιούν στο ίδιο μέρος. Και περίπου το ίμιση φτάνουν στο σύστημα αυτό μέσα από την Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, την Bundesbank. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ισολογισμοί του Target 2 αυξάνονται στη Γερμανία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, ότι η αγορά ομολόγων ε, δημιουργεί ε, μία βελτίωση σε ένα χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον όσον αφορά τους πολιτές των ομολόγων. Πρόσφατα μερικοί πούλησαν ομόλογα και αγόρασαν άλλες αξίες, όχι απαραίτητα εσωτερικές αξίες, ή προέβησαν σε άλλο είδους επενδύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ισολογισμοί target του βελτιώνονται. Target του balances. Ε, δεν ξέρω, ε, το 12 είχαμε τελείως διαφορετική εμπειρία. Πρέπει όμως να σας πω ότι δεν μοιάζει. Ή τότε τουλάχιστον το 2012 δεν υπήρχαν ενδείξεις κρίσης στο ευρώ που να αιτιολογούν αυτή την βελτίωση των target του balance. Ο κύριος Μαυρίδης. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά. ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, κοινή αγορά ή όχι, και ανεξάρτητα με το αν θα υπάρξουν αλλαγές μετά την εκλογή του κυρίου Τραμπ, νομίζω πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση ότι ορισμένα πράγματα στην Ευρωζώνη πρέπει να προχωρήσουν συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να σας υποβάλω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την Τραπεζική Ένωση. Όχι όμως για τον τρίτο πυλώνα. corporatives. Νομίζω ότι με βάση τις συνθήκες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν από το άρθρο 54 corporative, Είναι ομάδες, ένα είδος συντεχνίας με νομική υπόσταση που διαφέρει όμως από άλλους οικονομικούς φορείς. Είναι συντεχνίες με νομική υπόσταση, corporatives. Και... Όχι συντεχνίες, συνεταιρισμοί. Διαβάζω το άρθρο 54 της Συμφωνίας ε, Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ομάδα άλλους οικονομικούς φορείς. ή ε, νομικά πρόσωπα με ειδικέ ε, λειτουργικές αρχές που διαφέρουν από άλλους οικονομικούς φορείς. Η Τραπεζική Ένωση όσο έχει τώρα είναι τι μία είναι δίκαιη απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς. Αυτή αυτή η διαφορετική λειτουργία αναγνωρίζεται με κάποιο ε, πρακτικό τρόπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη, πέστε την γρήγορα. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με διαφορετικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με τους ε, κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία που αφορά σε προϋποθέσεις και όρους, άδικους όρους ε, που χρησιμοποιούν οι τράπεζες σε συμβόλαια που συνάπτονται. Κύριος Ντράγκη, ξεκινάμε με δεύτερη ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, Αυτό που ρωτήσετε εμπίπτει περισσότερο στην προστασία του καταναλωτή, δηλαδή να διασφαλίζει κανείς ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι δίκαιοι ε, όσον αφορά τους πελάτες των τραπεζών. Αν κατάλαβα καλά, αυτό που ρωτάτε εμπίπτει στις αρμοδιότητες εθνικών αρχών, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τώρα, το άλλο θέμα, το πρώτο σχετικά με τους ε, με τι εταιρείε αστικού εμπορικού δικαίου συνεταιρισμοί. Ε, οι συνεταιρισμοί κατά πόσο αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που προβλέπει η συνθήκη όχι. Αν είναι αυτή η ερώτηση, θα σας δώσω μισή απάντηση και θα σας πω ότι η εφαρμογή της αρχής της ε, προσθετικότητας έχει υγιείς ρίζες στην εποπτεία και στις ρυθμίσεις, στους κανόνες. Το άλλο μισό της ε, απάντησής μου θα πρέπει να σας το δώσω σε γραπτή μορφή γιατί η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ καλή και πρέπει να ελέγξω και εγώ την απάντηση που θα σας δώσω κατά πόσον θα είναι απόλυτα σωστή ή όχι. Κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες εάν ε, ισχύουν ε, αυτά που ρώτησε ο κύριος ε, ε, Φέρμπερ για το Target 2. Δεν κατάλαβα τι μας απαντήσατε. Ε, αν έχω σωστά στο μυαλό τα στοιχεία 2,8 δις ευρώ είναι τώρα ο, ο ισολογισμός σας. Μιλάμε για κρατικά χρέη, όχι μόνο στην Επιτροπή της Βασιλείας, αλλά και στην κοινή γνώμη. Τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, αν κρίνουμε από το Brexit, η προβληματική για τις ε, χρηματαγορές ε, είναι πιο σοβαρή στην Ιταλία, είναι πιο κοντά μας αυτό. Και 33% έχετε φτάσει στο όριό σας στην αγορά του χρέους. Πώς θα βγει η Ιταλία από την παγίδα αυτή του χρέους και ποιο θα αναλάβανε την ευθύνη. Γι' αυτό είναι πιο επίγον από το Brexit. Και δεύτερον, αν αυξηθούν τα επιτόκια στι ΗΠΑ, μήπω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να διατηρήσει τη σημερινή τη πορεία για τα επιτόκια. Όπως είπε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέρση, είπε πρόσφατα ότι μπορεί να ανατραπούν όσα προβλέπουν οι αναλυτές. Αν αυξηθεί το ε, δολάριο και συνεχίζει να πέφτει το ευρώ, πώς θα τα λύσουμε όλα αυτά και με ποια κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Uh, Πρώτον, απαντήσω στο πρώτο που ρωτήσατε. Έχουμε ένα πρόγραμμα εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού. Το ρίσκο το αναλαμβάνουν κατά 80% οι εθνικές κεντρικές τράπεζες κάθε φορά. Δηλαδή από αυτή την άποψη είναι προστατευμένη η ΕΚΤ κατά 80%. It's quite... Είναι σαφές, αρκετά σαφές, ότι για μακρά μια μακρά περίοδος με χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια και επανειλημμένα είναι γόνιμο έδαφος για κινδύνους ε, οικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που μπορεί να προέρθουν από άλλα ε, μεγάλα ξένα κράτη ε, αν αυξήσουν τα επιτόκια τους ή και από άλλες πηγές. Αυτό που μπορούμε εμείς να πούμε είναι ότι παρακολουθούμε αυτό το κίνδυνο πάρα πολύ στενά και πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε αυτό το ρίσκο και αυτό τον καιρό ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από την ε, ε, παρεμπόδιση της ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η ανάκαμψή μας να μην ε, εκτοξευθεί αλλά να αποτελματωθεί αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σήμερα για όρους ανάπτυξης. Ε, βέβαια, τούτο λεχθέντον δεν ε, αγνοούμε τον κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τους παράγοντες αυτούς και έχουμε και πριγνωσή των ε, επιπλοκών αυτής της κατάστασης μιας παρατεταμένης περίοδου επέκτασης και μεγάλης ρευστότητας. Ο κύριος Λάγκεν, διαβάζουμε για το Brexit ότι η Μεγάλη Βρετανία ενδεχομένως να επιδοθεί σε αθέμητο ανταγωνισμό στα φορολογικά. Αυτό έτσι και αλλιώς είναι τεράστιο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει αντιμέτωπο τα μικρά κράτη με τα μεγάλα. Αυτό πώς το αξιολογείται ως κίνδυνο του Brexit, ακόμα και αν είναι του απότερου ε, μέλλοντος. Κοιτάξτε, ναι. συχνά λέτε ότι έχουμε τόσο πολλές εξουσίες, τόσο πολλές αρμοδιότητες και είμαστε πανίσχυροι. Εφορία ακόμα δεν έχουμε γίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχουμε φορολογικές αρμοδιότητες. Δεν ρώτησα για το δικό σας κύρος και την αυθεντία σας. Την άποψή σας ρώτησα. Είναι κίνδυνος για την Ευρωζώνη και την οικονομική εξέλιξη. Ναι, αλλά πώς να το πω. αν εκφράσω την άποψή μου για αυτά τα θέματα σε άλλες χώρες θα μου πείτε ότι υπερβαίνω τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες μας. Δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό μας αυτό τον καιρό αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα μιλήσω ισπανικά. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω. Ερώτηση πρώτη για το Brexit. Τα είπαμε σχεδόν όλα αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να επιμείνω λίγο και στη συζήτηση που γίνεται για το fiscal stand της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, έχουμε το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, μάλλον πακέτο που εξήγηλε η Βρετανική κυβέρνηση για να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες του ενδεχόμενου Brexit ή να τις ε, αντικρούσει. Θα είναι μια όθηση φορολογική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή συνδέεται ή δεν συνδέεται με αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι εννοώ, σε ποιο βαθμό η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να φανεί υπερβολικά ισχνή δεδομένης φορολογικής όθησης που θέλουν να κάνουν τώρα οι Βρετανοί. Και μιλώ και για τη συναγματική ισοτιμία που θα επηρεαστεί. Δεύτερη ερώτηση αφορά την εκλογική νίκη του Τραμπ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Βράχει πρόθεσμα φαίνεται ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed, θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια και γρήγορα. Αλλά σε ένα χρόνο και λιγότερο θα υπάρξει και αλλαγή εκεί στην ηγεσία. Και μετά τις ε, δηλώσεις του επόμενου Προέδρου για ενδεχόμενη ανεξαρτησία της ΦΕΔ θα μπορούσε να ε, μας οδηγήσει στο ενδεχόμενο να είναι κάποιος ε, πιο εκεντρικός ε, εκεί κυβερνήτης, ο οποίος θα αυξήσει τα επιτόκια και αυτό θα είναι και εις βάρος του ευρώ και εις βάρος της ε, πολιτικής μας νομισματικής μέσω και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, on your first question, exactly... Ευχαριστώ. Ε, για την πρώτη σας ερώτηση, ποιο είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος, ο αντίκτυπος των ε, οικονομικών ε, σχεδίων του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωζώνη. Αυτό με ρωτάτε. Δεν έχω απόλυτη γνώση για να μπορώ να κάνω αξιολόγηση, αλλά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όσο σχετικό και αν είναι, όσο σχετική και αν είναι η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι πολύ μικρότερη η πραγματικότητά της από, την, από τόσα συμβαίνουν στην Ευρωζώνη. Βεβαίω θα έχει αντίκτυπο, αλλά καταρχάς δεν θα μπορούσα να τον αξιολογήσω αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, ο μέγεθος του, το μέγεθος του αντικτύπου θα περιοριστεί δεδομένων ακριβώ και των διαφορών στο μέγεθος των δύο οντοτήτων Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκής Ένωση. Και επίση σε σχέση με το πόσο ανησυχούμε για τι εξελίξει στο Ηνωμένο Βασίλειο και πώ αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη δική μας πραγματικότητα είναι ούτως ή άλλως θέματα που τα σκεφτόμαστε. Το άλλο ερώτημα που θέσατε για, την, για τα πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης, για την ΦΕΔ, για τον κυβερνήτη, το νέο ή το προσωπικό, δεν έχω απόλυτη γνώση, αλλά γενικώ να πω ότι αν υπονομευθεί η ε, ανεξαρτησία των κεντρικών ε, τραπεζών προφανώς δεν βοηθά αυτό κανέναν, κυρίως ε, ούτε καν την ε, κυβέρνηση στην επικράτη της οποίας βρίσκεται η τράπεζα που υπονομεύεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μόρισον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω είναι η Ιταλία. Και να συνεχίσω κάτι που ερώτησε και ο συνάδελφος Μπάλτ και ο κύριος Λάγκεν την επόμενη χρονιά ε, η Ιταλία θα πρέπει να επαναχρηματοδοτήσει 300 δις από το χρέο της. Αυτό είναι λόγος ανησυχίας για εμάς και για σας ως ε, κεντρικού τραπεζίτη. Και επίσης το επιτόκιο στο οποίο θα μπορέσει να επαναχρηματοδοτήσει η Ιταλία, αν είναι πάνω από 3% που είναι το μέσο, ε, ο μέσος όρος των όριμων ομολόγων, υπάρχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει. Και ε, το πρόγραμμα OMT θα μπορούσε να είναι κομμάτι αυτού του, αυτής της προσπάθειας. Από την Ιταλική κυβέρνηση έχετε δει α, βούληση να δεσμευθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό. Και ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω σύντομα είναι ε, η, ε, τα collateral shortages. Από την οικονομική κρίση και μετά είδαμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στις ασφάλειες ε, που δεν έχει όμως ε, ε, καλυφθεί από εξίσου υψηλό επίπεδο περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τις ασφάλειες αυτές και επίσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι κάνει για τη διάθεση, για τη διάθεση των κολάτερων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Για την Ιταλία, σαν να δώσατε τα, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε μου φάνηκε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω πολλά. Γενικώ η βιωσιμότητα του, ενός, του χρέους μιας χώρας ε, ουσιαστικά ε, ε, είναι αποτέλεσμα του κατά πόσο μπορεί να το πληρώσει το κράτος, της, το χρέος συγγνώμη, της Ιταλίας είναι βιώσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να το πληρώσει, Πρέπει να πω ότι η Ιταλία έχει από τα υψηλότερα πλεονάσματα, ε, πρωτογενή πλεονάσματα μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος δανεισμού έχει ομαλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Και η ανάπτυξη της Ιταλίας επίσης ανακάμπτει σταδιακά. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε στις ε, δάφνες μας. Ε, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό, ε, πολύ ψηλό χρέος στις, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οπότε είναι σημαντικό η χώρα να αρθεί στο ύψος και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στα πλαίσια του πακέτου σταθερότητας και ανάπτυξης για τα πλεονάσματα, αλλά και να επιμείνει στις προσπάθειες που κάνει για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίω ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, δούμε τι θα γίνει και με την ε, ανάπτυξη της Ιταλίας, έτσι ώστε αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της. Τούτου λεχθέντος, έχουν υπάρξει κάποια ενθαρρυντικά βήματα και σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική διακυβέρνηση και τον τραπεζικό ε, τομέα της χώρας. Έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, αλλά όπως ε, είπα και πριν, ε, δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Τώρα, στη ό,τι αφορά τις έχουμε ένα πλαίσιο κινδύνου για τις εγγύησεις, το οποίο αναθεωρούμε και νομίζω ότι έχει γίνει έχει γίνει αρκετά ε, συχνά η, η αναθεώρηση αυτή. Νομίζω ότι γίνεται άπαξ ετησίωση κάθε δύο χρόνια. Προς το παρόν θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι εν τάξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρτσος. Α, με συγχωρείτε. Ε, πάλι για το πρόγραμμα δανεισμού. Ε, για τις ε, εγγύσεις μου θέσατε ένα ερώτημα. Αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Τη προηγούμενης εβδομάδα ε, είδαμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, αλλά βεβαίω πάντα είναι τα θέματα αυτά στα χέρια των ε, εθνικών κεντρικών τραπεζών. Οπότε προ το παρόν αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα ε, και θεωρεί και το Διοικητικό Συμβούλιο ότι όντω είναι ανάγκη να γίνει αυτή η αναβάθμιση. Ο κύριο Κίτσος. Δύο ερωτήσει έχω. Στην Ελλάδα ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν βραχυπρόθεσμα μέτρα σε σχέση με το δημόσιο χρέος χώρας που θα μειώσουν περισσότερο το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους τα επόμενα έτη. Τα μέτρα αυτά θα είναι σε συμφωνία με την απόφαση του Eurogroup που ελήφθηκε το Μάιο του 2016. Από την άλλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε ένα περιβάλλον σταδιακά αυξηνόμενο κόστος εξυπηρέτησης μάλλον χρηματοδότησης ε, του χρέους ε, λόγω των εξελίξεων Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιο είδους πολιτικής αστάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα πρέπει να περιμένει η Ελλάδα ως βραχυπρόθεσμα μέτρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος μας. Και Πρόεδρε Ντράγκη, συνεχώς υπογραμμίζεται ότι για την νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται για να επιτύχει θα πρέπει αυτή να συνδυαστεί με μια επικοδομητική ε, ε, φορολογική πολιτική και πρόοδο σε ε, μεταρρυθμίσεις διαρθωτικές. Ωστόσο, πολλές ε, κυβερνήσεις έχουν ή κρίσιμες εκλογές ή μεγάλες πολιτικές δυσκολίες. Και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος του 2017 για να ανακαλύψουμε πόσα είναι εκείνα τα κράτη-μέλη που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν έτσι ώστε να διατυπωθεί και να εφαρμοστεί μια συνολική και αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Πιστεύετε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα μπορέσει να καλύψει το κενό που μόλις ε, περιέγραψα που θα προκύψει το ε, επόμενο έτος. Thank you. Well, uh, first thing is um, uh, Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξή. Αν δούμε λιγάκι τι συζητήσει που γίνονται ανάμεσα στου διάφορου αρμόδιου για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογή, είναι σαφέ ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ επιφυλάξει όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Έτσι λοιπόν είναι προς όφελος ε, της Ευρωζώνης, το σύνολό της, πόσο μάλλον της Ελλάδας, να αναζητηθεί μια ε, μακροπρόθεσμη, μακροχρόνια λύση που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους τόσο βράχη όσο και μακροπρόθεσμα. Στις 7 Νοεμβρίου στο Eurogroup ε, προετοιμάζονται προετοιμάστηκαν τα πρώτα μέτρα και ευελπιστούμε στο να συμφωνηθούν τα μέτρα αυτά ε, κατά την επόμενη συνάντηση. Εμείς λοιπόν προσβλέπουμε σε μία λύση η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει την πλήρη βιωσιμότητα ε, και του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριος Φον Βάιτσέκερ, κύριε Ντράγκη, δύο ερωτήσει έχω να σας υποβάλω. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το πρόγραμμα υποδομών του κύριου Τραμπ που ε, θα μπορούσε να είναι μια αχτίδα στην ε, ζωφερή κατάσταση μετά τις εκλογές της Ηνωμένης Πολιτείας. Η ΕΚΤ λέει ότι θα αυξηθεί η ανάπτυξη ο ΣΑ λέει ότι θα αυξηθεί η ανάπτυξη, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλα αυτά, ε, θα ελοπιθούν όλα αυτά που προβλέπει ο ΣΑ. Εγώ έχω να κάνω εξή ερώτηση. Η γερμανική κυβέρνηση με τις εκλογές ε, το 2017 ε, σκέπτεται αν εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα τότε ή ο, ο ΣΑ θα το επενέσει εξίσου και δεύτερον Πώς ακριβώς ε, εσείς ε, Πώς αξιολογείτε το ότι απέτυχε η ιδέα να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό συνταξιδοτικό ε, ταμείο. Και όσον αφορά και ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση με το πρόγραμμα των στρατηγικών επενδύσεων του 2.0, τι ακριβώς πιστεύετε από αυτόν. Εξάλλου, κατά την άποψή σας, ποια θα πρέπει να είναι η εξυγίανση που πρέπει να επικρατεί, θα πρέπει να επιταχυνθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο δανεισμός είναι περιβολικός ή θα πρέπει να υπάρξει μία καθυστέρηση και να δούμε τι θα κάνουν ακριβώς οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, πώς πρέπει να οργανωθεί η τι είσαστε υπέρ της εξυγίανσης με εθνικό πρόσημο ή υπέρ της εξυγίανσης με διεθνές πρόσημο. Να απαντήσω πρώτα στη δεύτερη ερώτησή σας. Είναι αλήθεια ότι η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Συστημικών Κινδύνων ε, έχουν δηλώσει ότι εξετάζουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν τα στοιχεία. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο ε, για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Υπάρχουν κάποια στοιχεία του τραπεζικού μας συστήματος όπου έχουμε πάρα πολλούς παίκτες αυτή βέβαια είναι πολύ αποτελεσματική, το κόστος είναι πολύ χαμηλό και αυτοί εξυπηρετούν πάρα πολύ καλά την οικονομία τους. Και υπάρχουν και άλλοι ε, ή άλλα, άλλες περιπτώσεις που ισχύει το αντίθετο, λίγοι παίκτες δηλαδή, ιδιαίτερα όμως αναποτελεσματικοί με πολύ ψηλό ε, κόστος, ε, πολύ ψηλό λόγο ε, εισόδων κινδύνου. Άρα δηλαδή όταν λέμε ότι ε, στην περίπτωση αυτή υπάρχει πράγματι κίνδυνος, πρέπει να δούμε τι ακριβώς εννοούμε. Και νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι ο τελικός στόχος είναι να υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να είναι και ισχυρό και ανθεκτικό αλλά να εξυπηρετεί εξίσου καλά την πραγματική οικονομία. Αυτές ε, θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές προσπαθώντας να σχεδιάσουμε μια ε, διαδικασία εξυγίανσης. Αυτά προς το πρώτο. Δεύτερον, το πώς θα γίνουν όλα αυτά δεν είναι απόλυτα σαφές. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνει κανείς όλα αυτά, δηλαδή για να επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε οποιοδήποτε κλάδο. Ένας τρόπος είναι να βασίζεται κανείς στην ατομική πρωτοβουλία, στα αυτοκίνητρα και στην δυνατότητα των ε, παραγόντων να βγουν τις καλύτερες συνέργειες, ε, τις καλύτερες προοπτικές και έτσι όλο αυτό αυτορυθμιζόμενο, ακριβώς επειδή υπάρχει και ίδιο συμφέρον, να καταλήξει κάπου στο βέλτιστο δυνατό σύστημα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι να υπάρχει έτσι ένας μεγαλεπίβολος ε, σχεδιασμός και αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι απόλυτα σαφές το τι θα κάνουμε. Γιατί δεν έχουμε σχεδιάσει το τι θα γίνει ακριβώς με τη δανειοδότηση. Και πάρα πολλοί στον τομέα της ε, νομοθεσίας είναι καινούργοι, δηλαδή Δεν είναι σαφές ότι τώρα επικρατεί ένα κλίμα το οποίο να στηρίζει την εξυγίανση. Το θέμα είναι να ορίσουμε τι είναι αυτό το overbanking. Πότε μπορεί να είναι αποτελεσματικό και πότε όχι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να υπάρχουν ε, ασαφείς σχεδιασμοί σχετικά με τον τραπεζικό τομέα. Το θέμα είναι πώς οι τράπεζες εξυπηρετούν τους πελάτες, ε, την πραγματική οικονομία και ποια είναι η λειτουργική τους, η επιχειρησιακή τους μάλλον αποτελεσματικότητα και θα πρέπει η εξυγίανση να γίνεται με βάση εθνικά πρότυπα ή όχι. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι απαραίτητο. Ίσως αυτό μερικές φορές πράγματι εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία, άλλες πάλι όχι. Αν θέλετε δεν βλέπω λόγους γιατί θα πρέπει να προβαίνουν σε εξυγίανση με βάση εθνικά πρότυπα. Δεν θα πρέπει αυτός ε, να είναι ο πρωταρχικός λόγος που θα επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Αυτά για την πρώτη σας ερώτηση. Για την δεύτερη είναι αλήθεια. Θα έλεγα ότι αν δούμε λιγάκι τις ε, δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί ουσιαστικά τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν οποτεδήποτε αυξάνονται οι δημόσιες επενδύσεις αυτό έχει θετικά συνεπακόλουθα και μπορεί να συμβάλλει ε, γενικότερα στην ανάπτυξη μιας χώρας γιατί κατ' ουσίαν αυξάνεται η κεφαλαιοποίηση και αν όλα αυτά είναι σωστά στοχευμένα πράγματι ε, βελτιώνουν, οδηγούν σε βελτίωση του αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η στόχευση, να υπάρχει καλή στόχευση. Γιατί ο λόγος που δεν είναι τόσο πολλές οι δημόσιες επενδύσεις είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις κατά παρελθόν οι επενδύσεις αυτές είναι απλά διασπάθηση. Πρέπει λοιπόν τις δημόσιες επενδύσεις να τις κατευθύνουμε προς εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες στηρίζουν την παραγωγικότητα και το δυναμικό ανάπτυξης. Και το έχω πει αυτό επανειλημμένα θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ε, να συστήσουμε τους εθνικούς μας προπολογισμού με τέτοιο τρόπο που να ε, κατευθύνονται περισσότερο σε φιλικό σχεδιασμό όπου μπορεί κανείς ε, να αυξήσει το σύνολο των κατακεφαλή δαπανών. Τώρα, όσον αφορά το FC2, Νομίζω είμαστε στο σωστό δρόμο. Αύξηση δημόσιων επενδύσεων, σωστά στοχευμένες επενδύσεις. Αυτό ε, θα αποβεί θετικό για το σύνολο της ευρωοικονομίας. Ευχαριστώ. Λούντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τράγκη. Ε, στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα καταλήξατε λέγοντας τα εξής. Η αντίδραση των αγορών, τον είπα, στην αρχή ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά μετά αμβλήθηκε και έδειξαν, είπατε, οι αγορές την ανθεκτικότητά τους. Και ε, ρωτώ, και οι τράπεζες γιατί γίνεται με την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, Bank of England και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, τα επαναλάβατε και σήμερα αυτά. Θα μπορούσατε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε. Ποιες είναι αυτές οι προετοιμασίες που κάνετε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι κάνατε πριν τις ε, Αμερικανικές εκλογές και μετά. Βεβαίως, η προετοιμασία ε, ε, το, της Bank of England και τη δική μας αφορά το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι την εκλογή Τραμπ προφανώς. είναι πολλές οι αλλαγές απλώς στις ε, τιμές ε, των στοιχείων ενεργητικού, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες μετά το δημοψήφισμα. Δεν φάνηκε να υπάρχει μεγάλη μετακίνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες έχουν γραμμές ρευστότητας. Επίσης εξασφαλίσαμε να ενισχυθεί η θέση τους, να υπάρχει αρκετή εποπτεία και ε, πριν το δημοψήφισμα, δηλαδή αν υπήρχαν κάποιες θέσεις που κινδύνευαν, ε, που ε, θα δημιουργούσαν ανησυχίες να αντιμετωπιστούν αμέσως. Τέτοιου είδους προετοιμασία κάναμε. Μάλιστα. Μια συμπληρωματική ερώτηση μόνο. Τώρα σταμάτησαν αυτά τα μέτρα ή προβλέπετε και άλλα τέτοιου τύπου. Τα θεωρείτε απαραίτητα στο προσεχές στο απότερο μέλλον. Όχι, δεν υπάρχει κανένα ειδικό μέτρο σε ό,τι μας αφορά σε να ενισχύουμε το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Ωραία, για ένα άλλο θέμα θέλω να ρωτήσω την 1η Νοεμβρίου είχα μια έκθεση της Deutsche Bank που έλεγε, μιλούσε για τη σκοτεινή πλευρά της ποσοτικής χαλάρωσης. The dark side of QE. Σωστά μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις. Λέτε και επιμένετε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και να τις υλοποιούν και στο έγγραφο αυτό της Deutsche Bank έλεγε ότι ακριβώς επειδή είναι χαλαρή η νομισματική σας πολιτική σταμάτησε αυτή η ε, φόρα που είχαν πάρει χώρες. Ας πούμε μέχρι το Ιούλιο του 2014 ήταν υψηλά τα επιτόκια και τα κράτη ήταν αγκασμένα να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Αν δείτε ε, τις ε, συστάσεις του 2012 μόνο οι μισές έχουν εφαρμοστεί ενώ του 2015 από τις συστάσεις μόνο το 1 πέμπτο. Δεν είναι καινούργια ερώτησή μου αλλά θέλω να την ξανακάνω. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση της Deutsche Bank συμφωνείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την παρέμβασή της φρέναρε κάπως αυτή τη φόρα που είχαν πάρει οι χώρες και έκαναν διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι τόσο ε, απαραίτητες όσο και επίγουσες ε, στα εργασιακά, στα κοινωνικά συστήματα, παντού. Απάντηση όχι, διαφωνώ. Επανελειμμένα έχω εξηγήσει αυτό το επιχείρημα δεν είναι προφανές ότι τα υψηλά επιτόκια κατά κάποιο τρόπο θα τόνωναν ε, το μεταρρυθμιστικό πνεύμα των ηθινόντων μας. Παράδειγμα, πρόσφατη εμπειρία. Είχαμε αλλαγές, σημαντικές ερθωτικές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά κυρίως και αλλού στην οικονομία, ενώ τα επιτόκια τα χαμηλά εδώ και καιρό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το εξή. Ας δούμε για ποιες διευθυντικές μεταρρυθμίσεις συζητούμε. Αν πιστεύουμε πραγματικά ότι συνδέεται το ύψος των επιτοκίων με τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, πιθανότατα εννοούμε μεταρρυθμίσεις που με κάποιο τρόπο έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός χρειάζεται χρηματοδότηση. Όσο πιο δύσκολη η χρηματοδότηση, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα εξορθολόγησης και εξηγίασή του. Ας πούμε, μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, όταν είναι τόσο σφιχτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτές, είναι αυτές άραγε οι διαστοτικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες κουβεντιάζουμε. Όχι προφανώς. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης, ας πούμε. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα. έχουμε μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, στον εκλογικό νόμο, στα συντάγματα. Πιστεύουμε σοβαρά ότι οι χώρες κάνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις όταν είναι υψηλά τα επιτόκια και δεν τις κάνουν όταν είναι χαμηλά. Αμφιβάλλω. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό. Και επίσης η έρευνα που κάνουμε εμείς στην ΕΚΤ δείχνουν ότι τα χαμηλά επιτόκια είναι κίνητρο για τις μεταρρυθμίσεις, γιατί οι μεταρρυθμίσεις συνήθως βλάπτουν κάποια συμφέροντα και ευνοούν κάποια άλλα. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι πόροι έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η ζημιά και να τονώνονται τα στρώματα εκείνα που έχουν τις μεγαλύτερες ζημίες. Δεν νομίζω ότι αφαιρέσαμε το κίνητρο με μία εξαίρεση αυτά τα πράγματα, ε, αυτά που συνδέονται με την χρηματοδότηση του προπολογισμού μιας χώρας. Ευχαριστώ. Μαρτουσέλο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ξαναπροσπαθήσω μία ερώτηση που έθεσε και ο Πρόεδρος κύριος Μπάλς. Πριν από λίγες μέρες οι Financial Times έγραφαν ότι αν έπρεπε να καταψηφιστεί το, ψηφοσμί, το δημοψήφισμα στην Ιταλία. Αν ήταν όχι, δηλαδή το αποτέλεσμα, θα έβγαινε η Ιταλία από το ευρώ. Εσεί πιστεύετε ότι μια χώρα μπορεί να βγει από το ευρώ χωρίς να το θέλει, απλά και μόνο επειδή θεωρεί ότι αυτό σημαίνει το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος Και το δεύτερο, μας είπε κάπως ο κ. Βάλλη, έδωσε κάποιες, κάποιους ε, Ιταλικές και αγγλικές εφημερίδες γράφουν με μη επιχαίους τίτλους ότι οκτώ Ιταλικές τράπεζες θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν όχι. Καταλαβαίνετε τώρα το πανικό, τον τρόμο του καταθέτη. Τι θα έκανε, θα έτρεχε γρήγορα γρήγορα ε, να πάρει τις καταθέσεις για να μην υπάρχει ο κίνδυνος του κουρέματος. Πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Bundesbank είναι ότι το πραγματικό πρόβλημα πρόβλημα είναι ότι οι πρόεδροι των κεντρικών τραπεζών είναι και πολιτικοί. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Περιμένουμε από εσάς ε, μία ένδειξη, εισαγωγικά ένδειξη πολιτική για να μας καθησυχάσετε. Να καθησυχάσετε τις αγορές και κυρίως τους καταθέτες. Γιατί σας λέω ειλικρινά, σήμερα οι πηχαίοι τίτλοι των εφημερίδων στην Ιταλία έχουν προκαλέσει αδίκως πανικό, τεράστιο πανικό και Ω εκ τούτου εγώ θεωρώ ότι αυτό απλά είναι άλλο εργαλείο για να εντείνουν τον διατραπεζικό ανταγωνισμό. Είπατε ότι δεν ξέρετε αν θα απαντήσω την ερώτηση. Δίκιο είχατε. Δεν θα απαντήσω. Εγώ λοιπόν δεν θα απαντήσω σε καμία από τις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο χρόνο για κάποιες έκτακτες ερωτήσεις. Ναι, αλλά δεν ζητήσατε συμπληρωματική ε, ερώτηση. Ε, ναι, ο, αυτός που θέλει να θέσει την ερώτηση πρέπει να, να τη ζητήσει. Δεν, δεν χρειάζεται δικηγόρο σας. Ορίστε, είναι έτοιμος λοιπόν ο συνάδελφος για τη συμπληρωματική του ερώτηση. Ε, Εντάξει, καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε την απάντησή σας, αλλά σας παρακαλώ πολύ, ε, έχετε κατά νου. Υπάρχει μια οικονομική εφημερίδα που λέει ότι αν ε, είναι όχι το αποτέλεσμα η Ιταλία θα βγει από το ευρώ. Ε, δώστε μου τουλάχιστον μια πάτση πάνω σε αυτό. Μπορεί μια χώρα να βγει από το ευρώ χωρίς να το θέλει απλά και μόνο επειδή η απάντηση του δημοψηφίσματος είναι όχι. Η ερώτηση, εντάξει, σίγουρα έχει σχέση με την εξαρτία που αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα στην Ιταλία. Καλύτερα αυτή να γίνεται στη δική μα τη χώρα. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τα σχόλια άλλων για τα άρθρα κάποιων τρίτων. Σα επαναλαμβάνω αυτό που σα είπα και πριν. Δεν θα πω τίποτα. Μάλιστα, κύριο Στόιρερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Πρόεδρε, Αναφερθήκατε στην ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Χρονικά μπορείτε να μας κάνετε ε, μία πρόβλεψη πόσο χρόνο έχουμε. Αν το ε, συγκρίνουμε τη ζώνη του δωραρίου με την Ευρωζώνη, διαπιστώνω ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες. Η διαφορά βρίσκεται στα πολιτικά όργανα και στις προσαρμογές. Άρα, δεν θα έπρεπε να είστε πιο σαφείς λέγοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες ε, μπορούν να επηρεάσουν τα βραχυπρόθεσμα ε, επιτόκια, ε, αλλά τα μακροπρόθεσμα εξαρτώνται από άλλους παράγοντες, κυρίως από τις προοπτικές ανάπτυξης. Και παρά την, το γεγονός ότι είναι χαμηλά τα επιτόκια, ιδιαίτερα στα ομόλογα, συνδέεται και με το γεγονός ότι οι διεθνείς χρηματαγορές ε, εκτιμούν ότι είναι χαμηλότερες οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Έχετε δίκιο. Πολλές φορές έχουμε πει ότι η νομισματική πολιτική αυτή που διευκολύνει πολύ θα οδηγήσει στην κυκλική ανάκαμψη. Αλλά για να είναι βιώσιμη αυτή η ανάκαμψη και μακροπρόθεσμα χρειάζονται και άλλες πολιτικές και κυρίως διαρθρωτικές πολιτικές οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το ε, δυναμικό που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Οπότε ως προς αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Η κυρία Μπερέσου. Κύριε Πρόεδρε, προφανώς θέλατε να πείτε περισσότερα για την έκθεση του ελεκτικού ε, συνεδρίου για τον ε, ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Ορίστε, σας δίνω την ευκαιρία να μας πείτε οριζοντίως και καθέτος τι πιστεύετε για το ελεκτικό συνέδριο που ανακατεύεται όλο και περισσότερο με την πολιτική και λιγότερο με λογαριασμούς, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να πω και πάλι ότι εκτιμούμε την έκθεση και ορισμένα από τα σημεία που αναφέρει και θέτει είναι πάρα πολύ χρήσιμο το γεγονός και μόνο ότι τα αναφέρει. Γιατί θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν θα ζητήσει θέματα στελέχωσης του ε, SSM. Ωστόσο, η έκθεση ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε πλήρης συνεργασία, λέει, από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και η δική μας εντύπωση είναι ότι έχουμε αφαιρώσει πάρα πολύ χρόνο στη συνεργασία μας με ε, την, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλλά η εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να ελέγχει ε, την ε, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, τα οικονομικά και όχι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεώρησει την εντολή του ελεκτικού συνεδρίου πολύ σύντομα. Το άλλο θέμα είναι ο διαχωρισμός. Δηλαδή, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, μοιράζονται κάποιες υπηρεσίες, όπως είναι η μηχανογράφηση, όπως είναι η ανθρώπινη πόρη και άλλα πράγματα. Αυτό ερμηνεύεται ως εναγκαλισμός και ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο διαχωρισμός είναι κατοχυρωμένος στην αρχή και είναι μια διάκριση ότι από τη μια έχει την εποπτεία και από την άλλη το, ε, την νομισματική πολιτική. Αυτές είναι μικτές ε, δραστηριότητες που δεν ε, έχουν να κάνουν ε, με το διαχωρισμό. Θέλουμε να αποφύγουμε τις πατάλες και τις επικαλύψεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδημόλης και ο κύριος Λάγκεν μετά. Herr Όχι, πρώτα ο κύριος Παπαδημόλης είπαμε. Thank you very welcome, Mr. Draghi. I'll speak in Greek. Uh, άκουσα με ενδιαφέρον την απάντησή σας στον συνάδελφο τον κύριο Κίρτσο ότι προσβλέπετε στην επόμενη ε, συνάντηση του Eurogroup σε μέτρα ελάφρυσης του χρέους, όπως είπατε επιλέξει και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και για το δημόσιο και για το ιδιωτικό. Ακούμε και δηλώσεις που λένε δεν χρειάζεται αυτό, δεν είναι καλό ούτε για την Ευρωζώνη ούτε για την Ελλάδα. Πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση για μετά από δύο χρόνια. Ποια είναι η απάντησή σας απέναντι σε αυτούς που λένε δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα γιατί δεν θα είναι ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρωζώνη καλό. Και επίσης πώς σχολιάζεται τη σημερινή ανακοίνωση του ΟΟΣΑ που λέει ότι απαιτείται πρόσθετη ελάφρυση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ε, κύριε Λάγκεν, κύριε Πρόεδρε, σωστά στο παρελθόν τονίσατε τις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Και σήμερα ψάχνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από πλευρά σας και έχω να ρωτήσω ε, κατά την άποψή σας ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στις τρεις, τρεις μεγαλύτερες χώρες του ευρώ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Ε, για να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Αν δούμε τώρα την κατάσταση, βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος από τον ελληνικό λαό τους τελευταίους μήνες. Και είναι πολύ σημαντικό να μην διαταράξουμε αυτή την πρόοδο. Το καλύτερο λοιπόν που μπορεί να γίνει τώρα είναι να υπάρξει επιτυχής ολοκλήρωση της, ε, ε, της αξιολόγησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην χάσουμε το χρονικό ορόσημο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ε, αξιολόγηση. Το δεύτερο τώρα ερώτημα, κύριε Λάγκεν, θέσατε πολύ δύσκολο ερώτημα. Κάθε χώρα έχει δικό της κατάλογο μεταρρυθμίσεων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει ένα φάσμα, ε, ανταγωνισμός, ε, υπηρεσίες, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς που και για τις τρεις χώρες επίσης θα αποτελούσε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί και στις τρεις χώρες. Επίσης, ε, η αγορά εργασίας. Ε, δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ε, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για την αναβάθμιση των ε, προσόντων των πολιτών για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσει της αγοράς. Είναι πολύ ευρύς λοιπόν ο κατάλογος αυτός μεταρρυθμίσεων, αλλά είναι και διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Με εξαίρεση βεβαίως την ενιαία αγορά. Η ενιαία αγορά είναι νομίζω διεθνικό σημείο. Ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο αυτό κομμάτι του νομισματικού διαλόγου και ο πρόεδρος Δράγκη θα επανέλθει σε λίγα λεπτά για το δεύτερο τμήμα ως ε, πρόεδρος της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Συστημικό Κίνδυνο. Οπότε θα προχωρήσουμε τώρα με την εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου. Διότι, όπως ξέρετε, ο Πάμπλο Ζάλμπα είναι ο πρόεδρος ε, του ε, Ινστιτούτου Credit Official. We let Pablo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 stay <laughs> Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον Παύλο Θάλμπα, όπως είπαμε. Ανέλαβε μια πάρα πολύ ε, σημαντική νέα θέση. Βεβαίως και θα μας λείψεις. Εξαιρετικός συνάδελφος, φίλος και πάρα πολύ καλός αντιπρόεδρος ήσουν. Και πραγματικά θα μας λείψεις αλλά δεν θα χαθούμε. Θα συνεργαζόμαστε μαζί ε, από τα νέα σου καθήκοντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Θερμότατα. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Μπάλτς. Εξ όσου γνωρίζω, Πρόεδρε, πρέπει να εκλέξουμε έναν τέταρτο αντιπρόεδρο στην Επιτροπή μας, αντικαταστάτη του κυρίου Θάλμπα, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θέλω να ε, προτείνω τον συνάδελφο Μάτο από την Ισπανία. Α, έπρεπε να έχω πει κάτι προηγουμένως όμως πριν πάρετε το λόγο. Ότι, εντάξει, με πρόλαβες. Ε, λοιπόν, τώρα θα πάμε στην εκλογή αντιπροέδρου και υπάρχουν και αντικαταστάτες ε, ε, μέλη ΣΠΑ που τα Γιάννη Μαν και Πρέντα θα ψηφίσουν. Είμαστε πάνω από 16 μέλη παρόντα. Έχουμε απαρτία. Yes. Μπορώ τώρα να προτείνω. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Όπως έλεγα, δυστυχώς θα πρέπει να αντικαταστήσουμε τον Παύλο ως τέταρτο αντιπρόεδρο διότι φεύγει και εξ ονόματο του ΕΛΚ προτείνω τον Καμπριέλ Μάτο από την Ισπανία για νέο τέταρτο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Συμφωνία ο υποψήφιος. Ναι. Ξέρω ότι είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής μας, τακτικό δηλαδή, και έχει υπογράψει κανονικά τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε διαβοήσει στην εκλογή του, αν συμφωνείτε. Παρακαλώ, ελάτε στο Προεδρείο. <laughs> Ωραία. Δύο λεπτά διακοπή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε. Έχουμε το δεύτερο μέρος τώρα της δημόσιας ακρόσης με τον κύριο Μάριο Τράγκη υπό την ιδιότητα τώρα ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που είναι αρμόδιος για τη μακρό ε, προληπτική εποπτεία. Την τελευταία φορά με την ιδιότητα αυτή ήρθε εδώ στις 23 Ιουνίου. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει εξελίξεις που αφορούν μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τράπεζες κτλ. Συστημικός κίνδυνος εκτιμήθηκε από το αντίστοιχο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και η ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης συστημικού κινδύνου εκδίδει κάποιες προειδοποιήσει τάσει. Θα τα ακούσουμε τώρα αμέσω από τον κύριο Ντράγκη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη τη οικονομική και νομισματική επιτροπή, κύριε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά έρχομαι να σας ενημερώσω για το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου επί την ιδιότητά μου ω Πρόεδρο. Από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε εκδώσαμε την ετήσια έκθεση που καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1η Απριλίου 2015 και 31η Μαρτίου 2016. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει ε, τις απόψεις μας για τον κίνδυνο και εξετάζει τη μακροπροληπτική ανάλυση, αλλά ταυτόχρονα δίνει μια εποπτεία των μέτρων που έχουμε λάβει στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις και τον αντίστοιχο κανονισμό και δίνει και συνέχεια ε, στα όσα έγιναν μετά τις προηγούμενες συστάσεις μας. Σήμερα όμως θα ήθελα να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα όσα μας είχατε αναθέσει να κάνουμε. Σχεδιάστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ως ανεξάρτητος φορέας ε, γενικότερα για το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αρκεί να δει κανείς τα μέλη συγκεντρώνονται κεντρικές τράπεζες, εποπτικές αρχές, ε, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή καθώς επίσης και ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί που εκπροσωπούνται στο Επιστημονικό Συμβούλιο, δηλαδή την αντίστοιχη επιτροπή. Είναι σημαντική αυτή η σύνθεση έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδυνού να ανταποκρίνεται στο έργο του γιατί δεν έχει δεσμευτικές εξουσίες. Είναι ε, ήπιος ο χαρακτήρας εξουσίας του και ε, συστάσεις μεταξύ ίσων. Θα ήθελα να σας αναφέρω τις πρόσφατες δραστηριότητες για να σας ε, περιγράψω τι κάνουμε για τις προτεραιότητες μας. Ε, σήμερα εκδίδουμε μια έκθεση ε, για θέματα χαμηλών επιτοκίων, διαρθρωτικών αλλαγών και ε, γενικότερα. Διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο ως φόρουμ συνεργασίας μεταξύ θεσμών που συνεισφέρει στη διαφύλαξη της οικονομικής σταθερότητας παντού στην Ένωση. Η έκθεση έχει εκδοθεί σε συνεργασία και με την Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή και ε, άλλες επιτροπές μας και είναι καταπληκτικό παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιστημικού Κινδύνου. Όταν συναντηθήκαμε για τελευταία φορά σας είχα πει ότι στόχος μας ήταν να εκτιμήσουμε το τι ε, σημαίνουν τα χαμηλά επιτόκια από συστημικής άποψης στην οικονομική σταθερότητα. Έχουμε μια συνολική προσέγγιση, καλύπτουμε όλους τους μεγάλους τομείς ε, στο σύστημα και βλέπουμε ε, πώς μπορεί να γίνει μεταφορά και μετάδοση από τον ένα τομέα στον άλλον όταν έχουμε συστημικό κίνδυνο. Είναι τρεις οι τομείς που έχουμε εντοπίσει. Πρώτον, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων. Δεύτερον, ε, η λήψη, η ανάληψη κινδύνου σε ευρεία βάση. Και τρίτον, οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με αλλαγές στη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε κάποιο βαθμό, η ανάληψη ε, κινδύνου ε, μπορεί να αυξηθεί ε, σε σχέση με τα επιτόκια όταν αυτά παραμένουν ε, ε, χαμηλά, αλλά υπάρχουν και πιο συγκυριακοί κίνδυνοι. Θα ήθελα σύντομα να σας αναλύσω τους τρεις τομείς που ανέφερα. Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, ένα περιβάλλον παρατεταμένων χαμηλών επιτοκίων πιέζει την κερδοφορία και την φερεγγιότητα των τραπεζών Ε, ας πούμε κάποιες ε, ε, μορφές ασφαλιών ζωής και συνταξιωτικών ταμείων έχουν εγγυημένη απόδοση και αυτό συμπιέζει το τραπεζικό τομέα και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητά του. Αυτό έχει να κάνει και με αρνητική επιρροή στην κερδοφορία τους γιατί είναι ασυμπίεστες οι καταθέσεις και χαμηλά τα επιτόκια. Ταυτόχρονα όταν παραμένει χαμηλή οικονομική ανάπτυξη δεν ε, μπορούν να αντισταθμιστούν οι απώλειες από δάνεια. Επιπλέον, δεν μπορούν ε, άλλες πηγές να ε, αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος. Επιπλέον, ο κίνδυνος οικονομικής σταθερότητας που συνδέεται με τις χρηματαγορές μπορεί να αυξηθεί όταν παραμένουν χαμηλά τα επιτόκια όταν κάποιοι ψάχνουν καλύτερη απόδοση. Όταν η μεγαλύτερη απόδοση αναζητείται σε μοχλεύση, ε, σε επισφαλή προϊόντα ε, και επίσης υπάρχει και κάποια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά κάποια βασικά στοιχεία ενεργητικού. Ε, μπορεί λοιπόν αυτός ο κίνδυνος να ε, επηρεάσει τους συμμετέχοντες στην αγορά και τους ισολογισμούς. Τέλος, τα χαμηλά επιτόκια ε, ενδέχεται να επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια δομή που να βασίζεται περισσότερο στην αγορά. Μετατοπίζονται οι δραστηριότητες στο μη τραπεζικό τομέα για να υπάρχει ένα είδος ρεζέρβας, ε, δηλαδή εναλλακτική πηγής χρηματοδότησης, εφόσον ε, δεν μπορούν οι τράπεζες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς στις τράπεζες και στις αγορές μεγαλύτερη ευαισθησία. Η έκθεση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου παρουσιάζει για κάποια μέτρα για να προλαμβάνονται όλα αυτά και να ε, περιορίζονται, να αμβλύνονται είναι σημαντικό να θεωρήσουμε τις πολιτικές μας από μια προοπτική ολιστική και σε όλο το σύστημα, ιδιαίτερα ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η κίνδυνη και η ανάγκη να περιοριστεί ε, το αρμπιτράζ. Γενικά, βασιζόμαστε στην αύξηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών, ε, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου της ανατίμησης ενίσχυση ε, του περιβάλλοντος και βελτίωση ε, του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά που συζητεί η έκθεση δεν θα πρέπει να τα αντιληφθούμε ως συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, αλλά μάλλον ως προτάσεις, έτσι ώστε οι αρμόδιοι και οι ενδιαφερόμενοι να συνεχίσουν τη συζήτηση. Ε, οι δυνατότητες πολιτικής περιλαμβάνουν μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν βράχη πρόθεσμα και όπου σε κάποιες περιπτώσεις ήδη συμπεριλαμβάνονται σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, υφιστάμενες ή και άλλα project που θα πρέπει ε, να εκτιμήσουν τον κίνδυνο και να τον περιορίσουν. Η έκθεσή μα επίση, τονίζει την ανάγκη να κλείσει το χάσμα δεδομένων που υπάρχει. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, οι κανονιστικές και ρυθμιστικές βελτίωσαν ε, τη χρήση δεδομένων και τη διάθεση δεδομένων ε, σε κάποιους τομείς του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, παραμένουν προβλήματα δεδομένων και θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία μεταξύ των τραπεζών με πλήρη χρήση ε, υφισταμένων πηγών δεδομένων ή μελλοντικών, όπως είναι το EMIR και το AIFMD. Ιδιαίτερα, οι απαιτήσει για αποκάλυψη και η μόχλευση ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουμε όλα αυτά υπόψη μας και με χαρά θέλω να σας πω ότι λαμβάνουμε ήδη ε, δράση για να μειωθεί αυτό το χάσμα των δεδομένων. Σήμερα ε, έχουμε μια σύσταση που καλύπτει ε, και τομείς real estate στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κτηματαγορά σε ορισμένες χώρες μέλη. Επιπλέον, το Συμβούλιο μας έχει ειδικέ ε, προειδοποιήσεις για 8 χώρες ε, στην κτηματαγορά ε, στον χώρο των κατοικιών. Ε, τα έχουμε ε, στείλει αυτά και στα 8 μελη στα αρμόδια υπουργεία. Έχουμε νομική εντολή να εκδίδουμε προειδοποιήσεις όταν υπάρχουν μεγάλη συστημικοί κίνδυνοι και να το επισημαίνουμε όταν χρειάζεται αυτό. Η ανάλυση μας είναι στραμμένη προς το μέλλον έτσι ώστε να βρούμε ποια είναι τα ευάλωτα σημεία και ο συστημικός κίνδυνος εγκαίρως έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζεται, να μετριάζεται αυτός ο κίνδυνος σε περίπτωση που υλοποιηθεί και υπέλθει δηλαδή πραγματικά. Ποια είναι τα βασικά ευάλωτα σημεία. Αυτά έχουν να κάνουν με τα χρεωμένα νοικοκυριά και ε, η δυνατότητα να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια. Επίσης, ε, ε, εκτιμούμε και πώς κυμαίνονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Η υπερχρέωση των οικοκυριών και η διακύμανση των αντικειμενικών αξιών χρειάζεται πολλά χρόνια μέχρι να οξυνθεί τόσο πολύ ώστε να δημιουργήσει ευάλωτες καταστάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να επέλθουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, ε, κόκκινα δάνεια, ε, μειωμένη κατανάλωση των οικοκυριών και ε, πτώση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 8 χώρε δεν είναι όλα τα ίδια. Και εμεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την κάθε χώρα. Παρόλο που γενικά τα ευάλωτα σημεία δεν συνδέονται με μεγάλο συστημικό κίνδυνο. Πρέπει πολύ γρήγορα να ληφθούν κάποια μέτρα γιατί η μακροπροληπτική ε, εποπτεία και άλλα μακροοικονομικά μέτρα ε, αποδίδουν περισσότερο όταν υιοθετούνται εγκαίρως. Τέλος, θέλω να πω ότι στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα εξακολουθεί να ασκεί ε, την εντολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εντοπίζει ακριβώς ζητήματα και ευάλωτα σημεία που έχουν να κάνουν και με χώρες. Έχει μια δομή θεσμική που του επιτρέπει να ασκεί πίεση μεταξύ ομοτήμων και να ε, αντιτίθεται ε, στην αδράνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να εντοπίζονται, να υπογραμμίζονται και να εκδίδουμε συστάσεις για άμεση δράση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, συνάδελφοι, να ξέρετε ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου. Τέσσερα λεπτά θα διερκει κάθε ερώτα απάντηση. Πρώτος ο κύριος Κίρτσος. 1,5 λεπτό. Η ερώτηση του, το, το μάγιστο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Έχετε να κάνετε και με συστημικούς κινδύνους που ε, είναι άσχετοι με τις τράπεζες και με τον σκιώδη περισσότερο τραπεζικό τομέα. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια ουσιαστική περιεκτική πολιτική για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους κίνδυνοι μη τραπεζική. Γιατί τόσο και οι δύο τομείς και ο τραπεζικός τομέας και ο σκιώδης τραπεζικός και οι δύο συνεχίζουν να εξελίσσονται. Αυτή η διαφοροποίηση σε μη τραπεζικό τομέα και σκιώδη τραπεζικό προσφέρει και ευκαιρίες αλλά και κινδύνους και πρέπει να ελέγχεται αυτή η εξέλιξη. Κίνδυνος είναι υπερβολική μόχλευση και επίση και υπερβολική συστημική αλληλένδεση η οποία υπάρχει κυρίως ανάμεσα σε πολλές ε, τράπεζες και τραπεζικά συστήματα και το πρόβλημα της ρευστότητας. Και αυτό απασχολεί κυρίως ε, τα μία που βασίζονται σε ομόλογα. Εμείς ε, λοιπόν τον πρώτη, την πρώτη υποπτία την, έχουμε, την κάναμε τον Ιούλιο του 2016 και αξιολογήσαμε τους κινδύνους κάτω από διάφορα πρίσματα. Πρώτον, μία προσέγγιση που αφορά στα διάφορα στοιχεία του ε, σκιώδους τραπεζικού τομέα συμπεριλαμβανομένου των ε, επενδυτικών ταμείων και πολλών άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στο μέλλον θα εξελίξουμε περαιτέρω το πλαίσιο ελέγχου της σκιώδους τραπεζικής αναλύοντας ε, διάφορα στοιχεία από το ΕΜΙΡ και επίσης και από την οδηγία AIFB, την εναλλακτική. Τώρα πόσο θα χρειαστούμε, πόσο καιρό. Όπως βλέπετε όλοι οι σημαντικοί φορείς σε αυτή την μικροπροληπτική, σε αυτό το μικροπροληπτικό εποπτικό περιβάλλον ε, για τον τραπεζικό και μη τραπεζικό τομέα. Αυτά υπάρχουν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να σα αναφέρω μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν ξέρω ακριβώ πότε, αλλά γνωρίζω ε, μια πολυετή διαδικασία και ως πρώην πρόεδρος ε, της EFSB ξέρω πολύ καλά πώς έχει αλλάξει το περιβάλλον και η νοοτροπία. Δηλαδή πλέον ε, είναι πολύ πιο ευνοϊκό το περιβάλλον στην εποπτεία, στο σχεδιασμό, ε, στο μικροπροληπτικό σχεδιασμό για τον τραπεζικό και μη τραπεζικό τομέα. Επειδή θα σας ανακοινώσω σύντομα πολύ ευχάριστα νέα σχετικά με τον ρυθμιστικό τομέα, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα. Η κυρία Περές. Ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον κύριο Ντράκη τη φρονή για τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης. Σε πάση εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό που λέει το πρόγραμμα εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προγραμματίζει αναθεώρηση του ε, θέματος τη διευκόλυνσης για την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Προς τα πού θέλετε να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε πάρα πολύ στην κτηματαγορά. Ε, στην αγορά κινήτων υπάρχουν ειδικοί τομείς όπου η εποπτεία του συστημικού κινδύνου δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένη από την ε, κείμενη νομοθεσία και από το σύστημα εποπτείας το οποίο έχουμε θεσπίσει και λειτουργεί. Στην αρχή επίση επιμείνατε στο γεγονός ότι δεν έχετε εκτελεστική εξουσία, δεν έχετε δεσμευτική ισχύ δηλαδή στα όσα λέτε. Αυτό τι σημαίνει. Υπάρχουν κάποιοι τομεί που πρέπει να αλλάξει νομοθεσία και να αποκτήσετε έτσι, ειδική εξουσία να παρεμβαίνετε. Έτσι, με δεσμευτική ισχύ, με υποχρεωτικό χαρακτήρα για να απαντήσω στο δεύτερο σας ερώτημα. Γενικώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρέχοντα σκοπό της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα ήταν ούτως ή άλλως ένας φορέας ε, λήψης αποφάσεων. Θα ήταν απλώς ένα φόρουμ, ένα βήμα, που, ένας φορέας που θα εκδίδει κάποιες συστάσεις, κάποιες προειδοποιήσεις, δηλαδή ένα ε, σημείο ήπιας ισχύω, όχι ένας φορέας δεσμευτικών, έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων, γιατί υπάρχουν άλλα θεσμικά όργανα που έχουν αυτές τις αντίστοιχες ακριβώς ε, αρμοδιότητες και σε εθνικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλοί φορείς που έχουν δυνατότητα έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου νομίζω ότι ε, με πολύ ικανοποιητικό, ικανοποιητικό τρόπο έρεται στο ύψος των καθηκόντων του. Τώρα, ο βασικός ε, κίνδυνος αυτή τη στιγμή, ο βασικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή, και παραλαμβάνω κάτι που είπα πιο πριν, είναι ε, να υπάρξει ε, στασιμότητα ή ε, παρεμπόδιση της ανάπτυξης και αυτό βεβαίως μεταφράζεται σε, οικονομικ... σε κινδύνους οικονομικής σταθερότητας. Αυτό είναι το σημείο κλειδί που πρέπει να έχουμε σήμερα υπόψη μας. Πιο συγκεκριμένα, ως... Έχουμε το θέμα της αποδυνάμωσης των, ασφαλιών, των ασφαλιών, των ιδρυμάτων, των ισολογισμών των τραπεζών και ο δεύτερος κίνδυνος είναι η ανατίμηση των, ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Βεβαίως θα υπάρξει μια τέτοια αναδιάρθρωση, αλλά θα είναι μάλλον ε, τραυματική. Ε, τρίτος κίνδυνος είναι η υποβάθμιση της βιωσιμότητας του χρέους και, στην, και στο κρατικό επίπεδο και στο επίπεδο των οικοκυριών. Και επίσης ο κίνδυνος μετάδοσης από τον σκιώδη τραπεζικό τομέα στον στο οικονομικό σύστημα. Αυτή είναι κίνδυνοι που δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητο ότι θα γίνουν, αλλά είναι ενδυνάμει κίνδυνοι ε, στους οποίους πρέπει να στρέψουμε την ε, προσοχή μας. Ευχαριστώ. Σάντερ Λούνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, την Πέμπτη είδαμε ότι οι μέτοχοι της ε, Banca Monte dei Paschi ενέκριναν ε, την έκδοση ε, ε, μετοχών ύψους 5 εκατομμυρίων. Πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό μέχρι το τέλος του έτους, μετά το stress βεβαίως που στο οποίο επιβλήθη η τράπεζα και είδαμε ότι είναι πιο αδύναμη, οπότε από εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Το σχέδιο αυτό θα, συνεχιστεί με την βοήθεια κάποιων ιδιωτικών ας πούμε, πρωτοβουλειών και επενδύσεων έχει πέσει το απόθεμα κατά 90% από το 2009. Οπότε το ερώτημα είναι, το σχέδιο αυτό θα πείσει, θα ελκύσει τους ε, επενδυτές. Και δεύτερο, πιο γενικό, ερώτημα, ο ίδιο σκεπτικό ωστόσο. Θεωρείτε ότι οι ε, λύσει με βάση την αγορά για τις ε, ε, σε κίνδυνο βρισκόμενες Ιταλικέ τράπεζε θα αρκέσει για να αντιμετωπίσει την, το πρόβλημα, την κρίση στον τραπεζικό κλάδο ή η Ιταλία χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό. Και τελευταίο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετίζεται και με το δημοψήφισμα που θα γίνει στην Ιταλία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου μελετά τον κίνδυνο, τον αντίκτυπο στη, στον τραπεζικό τομέα μιας ε, αρνητικής απάντησης στο δημοψήφισμα. Έχετε σκεφτεί κάποια έτσι ίσως ε, αρνητικά σενάρια που προκύψουν Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα λέγοντας ότι δεν σχολιάζω επιμέρους μεμονωμένα θεσμικά όργανα. Για το δεύτερο ερώτημά σας, όχι. Πόσο ξέρω τουλάχιστον. Οπότε, ε, μας μένει το άλλο σας ερώτημα, όπου ρωτάτε αν οι αγορές, οι λύσεις με βάση ε, την αγορά μπορούν να βοηθήσουν. Με βάση το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι, αγο, οι λύσεις επί της αγοράς πρέπει να είναι οι πρώτες που έρχονται ε, σε διερεύνηση όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σομπό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη που ήρθατε για άλλη μια φορά να μας βοηθήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να πάω λίγο στη ρίζα όλων αυτών που μας περιγράψατε. Ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου είναι μία λέσχη συζητήσεων, ε, συστάσεων, ε, συμβουλών και ότι δεν χρειάζεται εκτελεστική εξουσία. Είναι γεγονός και μπορεί να είναι η άποψή σα. Αλλά στην ουσία τι γίνεται. Δίνει πολύ την εντύπωση ότι συνεχίζει ο συστημικός κίνδυνος να είναι τέτοιος γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα να μεταρρυθμιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και υπάρχει το θέμα του too big to fail ή του interconnected to fail. Οπότε κάποιοι μεγάλοι προστατεύονται. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πηγές κινδύνου που συνδέονται με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Και τίποτα δεν ε, εξασφαλίζει ε, τους ε, πολίτες και την αγορά για το ότι κάνουν τα stress test και ποικίλει ε, η μεθοδολογία ανάλογα με την τράπεζα, αν είναι περιφερειακή, ανάλογα με τη χώρα, αν είναι ταμιευτήριο ή περιφερειακή τράπεζα. Και δεν μιλώ για το ιταλικό πρόβλημα που ακούσαμε προηγουμένω. Αυτά, εντάξει, αυτά, Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράκη. Thank you. Um, on... Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση. Έχουν ήδη γίνει πολλά Γιάννη, με το, το πιστεύω κίνδυνο του too big to fail. Ότι είσαι πολύ μεγάλος για να απτοχεύσεις. Αν δούμε τι έγινε λίγα χρόνια πριν την κρίση, οι δείκτες ε, κεφαλαίκοι ήταν 7% για την Ευρωζώνη, τώρα είναι 14%. Ε, υπάρχουν διάφορα μαξιλαράκια, buffer και προστατευτικά που έχουν γίνει, ιδιαίτερα και υποπτία παντού για την Ευρωζώνη αλλά και γενικότερα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ε, θεσπιστεί και τώρα για ε, το big to fail, έχουμε μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων. Έχουν γίνει πολλά. Είναι αρκετά αυτά, άρα ε, θα δείξει. Ο στόχος ποιος είναι. Για κάθε εποπτικό ή κανονιστικό πλαίσιο. Στόχος δεν είναι να είναι όλα ε, αεροστεγή για την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση, γιατί δεν ξέρουμε από πού θα προέλθει. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο στιβαρό και ανθεκτικό το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα μας. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας για τα stress και το σύστημα ΣΡΕΠ e ότι εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο, ομοιόμορφα αρκετά εφαρμόζεται αυτό σύμφωνα με τους ε, γενικούς και ε, ειδικούς κανονικούς κανόνες. Καλά, μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη και εγώ δεν είμαι αντικειμενικό όταν λέω αυτά, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα ε, αυτό το σύστημα των δοκιμών το Ο Κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Please use your headphones, Mr. Draghi. I will speak in Greek. Ε, κύριε Ντράγκη, υπάρχει εκκρεμότητα εδώ και χρόνια στην ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης και στη δημιουργία του περίφημου τρίτου πυλώνα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, το περίφημο σύστημα EDIS. Έχει κατατεθεί μια πρόταση της Κομισιόν με ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησης μέχρι το 2024. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη της, τη δική σας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αυτό τον τρίτο πυλώνα, γιατί το συζητούμε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πολλοί θεωρούν ότι χωρίς τον τρίτο πυλώνα δεν ολοκληρώνεται η τραπεζική ενοποίηση και παραμένουν σοβαροί συστημικοί κίνδυνοι που μεγαλώνουν. Ποια είναι η δική σας γνώμη από αυτού. Η απόψή μα είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο τρίτο πυλώνα για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και έχουμε την αίσθηση ότι η μείωση του κινδύνου θα πρέπει να συμβαδίζει χέρι-χέρι με την ε, μοιρασιά του κινδύνου. Δηλαδή, ε, έχουν γίνει πολλά για να μειωθεί ο κίνδυνο, το risk reduction, ε, ο επιμερισμό, α πούμε, ε, ανέφερα προηγουμένως τα διάφορα buffer το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για ε, την έκθεση, ε, αλλά όλα αυτά είναι σταδιακά, είναι μια διαδικασία. Το γνωρίζουμε αυτό και δεν είναι επίμαχο το θέμα, αλλά ειλικρινά έχει σημασία. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι γεγονός ότι οι σημερινές προτεραιότητες τα μυαλά των ηγετών μας φαίνεται να έχουν μετατοπιστεί για, σε πιο πιεστικές ανάγκες είναι στραμμένοι και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι ένας καλός λόγος να ξεχάσουμε όλα αυτά που είναι σημαντικά και παραμένουν. Και για να ολοκληρωθεί και να αντιμετωπίσουμε ε, τη, θα ευάλω τα σημεία, θα πρέπει να συμπληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, να γίνει η Ένωση Κεφαλαιογορών και αυτός είναι ένας πυλώνας. Ευχαριστώ. Η Μόλι Σκοτ Κέιτο. Όχι, αποσιάζει. Ο Ντέιβιτ Κόμπορν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι κύριε Ντράκη που σας ξαναβλέπω. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε την ε, κατάθεση ενός whistleblower σχετικά με τη Unicredit στην Ιρλανδία και διερωτώ με, αυτά τα ξέρατε όταν εσείς ήσταν τότε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ιταλικής Τράπεζας ή μήπως σας το απέκρυψαν. Οι ε, Ιρλανδοί ενημέρωσαν τους Ιταλούς και αν όχι γιατί όχι. Αυτά μας ανησυχούν κάτω από το κίνδυνο του συστημικού κινδύνου. Ε, η Unicredit είναι μία από τις μεγαλύτερες Ιταλικές τράπεζες. Δεν ξέρω, έχετε να πείτε κάτι από αυτού, να μας ενημερώσετε. Uh, ε, στην τελευταία συνεδρίαση στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, απάντησα ακριβώς αυτή την ερώτηση που είχε ε, κάνει ο κύριος Φλάναγκαν, αν δεν απατώμε. Και θέλω να σας πω ότι είχε προετοιμαστεί μια γραπτή απάντηση και ε, θα του σταλεί όπως ε, πάντα κάνουμε. Δεν ρώτησα αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να τη στείλετε και σε εμάς, ίσως και σε μένα. Με ενδιαφέρει να τη δω. Μας ανησυχεί πολύ. Γιατί θα πρέπει να τις προσέχετε. Έχουν υπερβολική υπερεξουσίες οι τράπεζες. Και είναι πάρα πολύ συχνά στις ειδήσει και στα πρωτοσέλιδα οι τράπεζες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει εσείς να εξασφαλίσετε ότι λειτουργεί σωστά το σύστημα. Και πολλοί εδώ θα ήθελα να ε, μάθουν περισσότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου στείλετε την απάντηση. Ευχαριστώ. κύριος Άνεμας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια αναθεώρηση αυτόν τον καιρό για το Macro Prudential ε, ε, Policy Framework στις 7 Νοεμβρίου συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε ένα briefing στις 22 Νοεμβρίου ε, τα δημοσίευσε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν άκουσα καλά και διάβασα καλά, θα εκχωρηθούν εθνικές αρμοδιότητες σε υπερεθνικό επίπεδο. Βέβαια αυτό δεν το έλεγαν με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, ήταν πιο διπλωματική και πιο συγκαλυμμένη η διατύπωση. Αλλά ποια είναι η σωστή ισορροπία, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πώς θα πάρετε εθνικές αρμοδιότητες. Αυτό μπορεί να σημαίνει streamlining, λέει, τα εργαλεία και ενισχύει το ε, ρόλο του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου στα πλαίσια ε, της λειτουργίας του SSM και ρωτώ Αυτή είναι μια εκχώρηση αρμοδιοτήτων υποβόσχουσα και υπόγεια και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σφετερίζεται τις ε, αρχές των εθνικών ε, ρυθμιστών. Αυτά τα θέματα ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι θα κάνει τώρα, θα εκχωρήσουμε σε κεντρικό επίπεδο και άλλες εξουσίες, εξουσίες που κανονικά ρυθμίζονται και ελέγχονται πολύ καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να σας πω. Ε, αυτό που έχει απαντήσει το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου μπορώ να σας πω. Αυτό που απάντησε στην Κομισιόν. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να υπογραμμίσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, και λέμε ότι το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αρμοδιο... Ε, εξουσιών από ένα επίπεδο σε άλλο. Είπαμε επίσης ότι ε, το Συμβούλιο ε, θα συνεχίσει να έχει την ευρεία του σύνθεση σύμφωνα και με την ε, λειτουργία που έχει από την, από την εντολή του να συγκερνά εμπειρογνώμονες από διάφορα θεσμικά όργανα. Αυτό πάλι δεν έχει να κάνει με μεταφορά εξουσιών. Μιλούμε για την απλούστευση της διαδικασίας ενεργοποίησης, για τα εργαλεία, για τον τραπεζικό τομέα. Και εδώ έχουμε κάνει μια γνωμοδότηση. Δεν, πάλι δεν μιλάμε για μεταφορά ε, εξουσιών, ε, εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Οπότε αυτά είναι τα θέματα που είχαμε, μας είχαν θέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτές τις απαντήσεις δώσαμε. Μετά, Είπαμε ότι τα μακροπροληπτικά εργαλεία εκτός του τραπεζικού τομέα υπάρχουν για συγκεκριμένους ε, λόγους, αλλά υπάρχει μια γενική ανάγκη να υπάρξει ένα ε, συνολικό, μια συνολική εργαλειοθήκη μακροπροληπτικών εργαλείων. Ε, για το μη τραπεζικός τομέας και ο σκιώδης τραπεζικός τομέας αυξάνονται πολύ γρήγορα και πρέπει να έχουμε μια εργαλειοθήκη στα χέρια μας για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια μακροπροληπτικά μέτρα για να μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ποιο θα το εφαρμόσει βεβαίω αυτό το πλαίσιο ακόμα είναι εκρεμέ. Θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι οι Εθνικέ Αρμόδιε Αρχέ. Ε, δεν έχουμε ε, απάντηση ακόμη στο ερώτημα αυτό. Άρα, συμπληρωματική ερώτηση. Υποθέτω ότι εσείς δεν παίξατε κανένα ρόλο στη συζήτηση αυτή τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς προσωπικά δεν παίξατε καθόλου ρόλο. Παίξαμε το ρόλο που μας ε, ανέθεσε η ερώτηση του Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτή την ερώτηση απαντήσαμε. Ε, Τέσσερα λεπτά έχουμε πει, παρεμβαίνει ο Πρόεδρος. Είσαστε πολύ αυστηρός κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ε, ε, ερωτήσεις ε, για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Τόμασμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γερμανικά, κύριε Ντράγκη. Η εντολή στην οποία αναφερθήκατε να κάνετε προειδοποιήσεις για συστημικό κίνδυνο. Αυτό δεν είναι μόνο αλλά μπορεί και να μας βοηθήσει, αλλά κανείς δεν είναι νησί. Δηλαδή, είναι κοινή ευθύνη και συνολική. Και σας ερωτώ, στο Brexit ήδη στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο ε, άρχισαν να υπάρχουν κάποιες διακοιμάσεις και μετά από αυτή την ε, ε εκλογή έκπληξη στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, έχουμε νέα δεδομένα. Μιλήσατε για την αγορά ακινήτων. Έχουμε ένα μεγιστάνα των ακινήτων, τον κύριο Ντόναλτ Τραμπ που είναι τώρα πρόεδρος των ΗΠΑ και θέλει να ακυρώσει διάφορες εμπορικές συμφωνίες, να τις αναστείλει, τι άλλες. Και μπορεί να υπάρξει αρνητική εξέλιξη. Δεν έχουμε πια εκείνη τη δυναμική της ανάπτυξης που αναφερθήκατε προηγουμένως αν αυξηθούν τα επιτόκια ή αν αυξηθεί ακόμα το κρατικό χρέος των ΗΠΑ ή ε, τι θα γίνει με τις τράπεζες. Μπορεί εμείς ε, να τις έχουμε σε κάποιο έλεγχο και σε κάποια ρέγουλα στην Ευρώπη και τις σκιώδεις και το μη τραπεζικό τομέα. Η Αμερική όχι. Αυτή η αύξηση του προστατευτισμού μήπως είναι μεγάλος κίνδυνος να αλλάξει η οικονομική μας ατζέντα, το πρόγραμμά μας. Μήπως είναι κίνδυνος για την οικονομική σταθερότητα για μας, την Ευρωζώνη και τη χρηματοπιστωτική. Δεν είναι εύκολο να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, γιατί θα σήμαινε ότι πρέπει να κάνουμε υποθέσεις για πολιτικές που ακόμη δεν υπάρχουν. Αυτές οι πολιτικές ε, αποτελούν ε, αποτέλεσμα εκλογικών ε, εξαρτιών, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη σε φάση σαφούς δήλωσης για το τι θα σημάνει αυτή η πολιτική για, την επόμενη, για τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε και μπορούμε να πούμε ότι ο προστατευτισμός δεν αυξάνει την ευημερία. Δεν αυξάνει την ευημερία των πολιτών. Και μετά πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει αυτό το κύμα προστατευτισμού. Μία από τις απαντήσεις είναι ότι έχουμε αγκαλιάσει την ε, παγκοσμιοποίηση τόσο πολύ, χωρίς όμως να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ζημιώθηκαν τελικά από την ε, ε, παγκοσμιοποίηση. Και ήταν πολύ παντού στον κόσμο. Το δίδαγμα λοιπόν που μπορούμε να αντλήσουμε τώρα είναι όχι να πάμε πίσω σε κάτι που ούτως ή άλλως ήταν αδύνατο να, να, να πάμε πίσω μέσω του προστατευτισμού, αλλά να φροντίσουμε πλέον αυτούς που έχουν χάσει πολλά Ακριβώ λόγω τη όλη διαδικασία τη παγκοσμιοποίηση χωρί φυσικά να ακυρώσουμε τα ωφέλη που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση τα τελευταία 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Πολ Τάγκ. Uh, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα. Ε, ε, έχουμε κάνει πολλές ε, συζητήσεις στο Κοινοβούλιο Είχαμε πει ότι πρέπει να λύσουμε διάφορα διδάγματα από την κρίση. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες εντός του Κοινοβουλίου για το... Ε, την τιτλοποίηση και πώς ε, ε, μπορεί να δημιουργήσει ίσως ε, τις διάφορες φούσκες που προκύπτουν από καιρούς καιρών θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η άποψή σας, αν κατανοείτε αυτές τις ανησυχίες που έχουμε, αν θεωρείτε ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου να παίξει κάποιο ρόλο στο να αμβληνθούν λίγο αυτές οι ανησυχίες, γιατί προς το παρόν για μας είναι δύσκολο να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση που θα προκύψει, αλλά ίσως το Συμβούλιο σας να μπορεί καλύτερα να εποπτεύσει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Το γεγονός είναι ότι ε, η τιτλοποίηση είναι ως τιτλοποίηση μάλλον αποκαλέσαμε διάφορα στοιχεία που ήταν τελείως διαφορετικά. Τιτλοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τιτλοποίηση στις ΕΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα subprimes, όταν ε, αυτά αποτέλεσαν ε, αποτέλεσμα αυτής της τιτλοποίησης, είτε ήταν πολύ δύσκολο κολλά συστήματα στην τιμολόγηση, ε, με τα λάθος κίνητρα στη φορά το κίνδυνο γιατί οι τράπεζες δεν ε, ε, ανέλαβαν καθόλου κίνδυνο η δική μας ε, ήταν τελείως διαφορετική από αυτό ήταν πιο διαφανής είχε αρκετή ορατότητα υπήρχε καλή τιμολόγηση και αυτό που φαίνεται είναι ότι ο, ο ρυθμός των ε, πτωχεύσεων ε, από τις ΙΠΑ ε, είναι πολύ πιο υψηλός από το δικό μας. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά τουλάχιστον τα δικά μας τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πολύ χαμηλά. Και παρόλα αυτά, η διδλοποίηση, αν σχεδιαστεί σωστά, είναι πολύ ισχυρό εργαλείο για την επέκταση των πιστώσεων και για την πραγματική οικονομία και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εντός λοιπόν αυτού του σύμπαντος, όπου ήδη υπάρχει ένα αρκετά αποδεκτό ε, προϊόν τυπλοποίησης, ε, μπορεί όντως να δημιουργηθούν ε, κάποιοι ακόμη κίνδυνοι. Κατά την άποψή μας λοιπόν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή ε, ο κίνδυνος ε, διακράτηση, ε, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι είναι, έχει μια καλή ισότητα γιατί αφήνει την αγορά να εξελιχθεί αλλά διατηρεί και έναν κίνδυνο και μια, ένα βαθμό πρόληψης. Τούτου τελευταίου βεβαίω είναι και τα επιτόκια πολύ χαμηλά οπότε δεν πρόκειται να δούμε μεγάλη ανάπτυξη του, του, του εργαλείου, τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμη, γιατί κάτι από αυτά που μας απασχολούν πέραν των περιορισμένων απολειών στην Ευρώπη, αυτό που έχουμε δει είναι να καταραίει η αγορά. Που, και η αγορά που κατέρευσε δεν ανέκαμψε. Δεν βοήθησε λοιπόν την σταθερότητα καθόλου αυτό. Ε, εντάξει, δεν ε, μπορούμε πάντα να συγκρίνουμε με τη ΣΥΠΑ, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ρόλο να παίξει έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή, στέρεη αγορά και να υπάρχει ρευστότητα όχι μόνο στους καλούς καιρούς αλλά και στους δύσκολους. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν η τιτλοποίηση σχεδιαστεί σωστά ως δυνατότητα διακράτησης κινδύνου, νομίζω ότι μπορεί να ε, αντιμετωπίσει και την ροή των ε, πιστώσεων για να μπορέσουν ε, τα δάνεια να φτάσουν στην πραγματική οικονομία. Είναι θετική συμβολή, εάν σχεδιαστεί σωστά. Για να υπάρξει ανάκαμψη της αγοράς βεβαίως θα πρέπει κατά αναγκή να υπάρξουν πιο υψηλά επιτόκια και επίσης να υπάρξουν ρυθμιστικές αλλαγές για τούτη την αγορά. Γιατί με τους παλαιότερους κανονισμούς καταφέραμε να, δούμε τα, να διαχειριστούμε τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά προϊόντα με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που ήταν τελείως διαφορετικά προϊόντα. Οπότε, αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό αξίζει τον κόπο, πρέπει να προσαρμοστείτε. Ευχαριστώ. We μπορούμε λοιπόν τώρα πλέον να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντράγκη. Ευχαριστούμε πολύ που με την ιδιότητά σας ε, του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου θα είσαστε πάλι εδώ το Μάιο του 2017. Βέβαια με την ιδιότητά σας του Προέδρου της ΕΚΤ φαντάζομαι ότι θα σας δούμε πολύ νωρίτερα. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα δύο λεπτών.

Λοιπόν, συναδελφοί, προχωράμε ε, με τη μισή διάταξη. Περνάμε στι ανακοινώσει του Πρόεδρου. Ενημέρωση για το συνεχιζόμενο τριμερή διάλογο. Δεύτερος διάλογος για τον κανονισμό προσπέκτους έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου. Ε, καλύψαμε τις εξαιρέσεις, ε, την έγκριση του κανονισμού, τη δημοσίευση του προσπέκτους, ε, στοιχεία τρίτων χωρών. Η πρόοδος ε, σημειώθηκε σε ορισμένα θέματα και ο επόμενος ημερής διάλογος προβλέπεται κατ' ουσίαν για αύριο. Όσον αφορά τα ταμεία των αγορών, Πρέπει να σας πω ότι επιτεύχθηκε συμφωνία στις 14 Νοεμβρίου στον 5ο τριμερή διάλογο μετά τις διαπραγματεύσεις που είχαν διαρκέσει από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβρη. Και αυτή η συμφωνία προβλέπει τρία, τρεις μορφές ε, τέτοιου είδους ε, ταμείων που προβλέπονται και αυτά ε, στους κανονισμούς. Αυτά τα τρία ε, ταμεία που σας ανέφερα ε, θα υπάγονται στις διατάξεις ε, διαφάνειας και ρευστότητας και θα υπάρξει κυρίως μια επιπρόσθετη πρόβλεψη το νέο πλαίσιο προβλέπει τα ταμεία αυτά να είναι πιο ανθεκτικά σε περίοδο κινδύνων. Επίσης έγινε και η τεχνική δουλειά του τριμερούς διαλόγου. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε έλεγχο, σε τελικό έλεγχο από τα διαπραγματευόμενα μέρη και η Επιτροπή θα επανέλθει εν ευθέτω χρόνο. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα λάβει χώρα κατά το ε, πρώτο τρίμηνο του 2017. Θέλω λοιπόν να ε, συγχαρώ την Νίνα Γκέιλ ε, και όλους ε, τους υπόλοιπους που συμμετείχαν σε πραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Η Κοινή Επιτροπή του, της Επιτροπής Προλογισμών και της ΕΚΟΝ αναβλήθηκε. Θα συζητηθεί το θέμα του προπολογισμού 13 Νοεμβρίου ήταν να λάβει η χώρα, τώρα θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου. Η ώρα της συνάντησης θα σας ανακοινωθεί σύντομα. έκον και Λίμπε, οι δύο αυτές επιτροπές θα συνεδριάσουν από κοινού 5η, 1η Δεκεμβρίου από τις 8 το πρωί στις 9 θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεσης ε, ε, για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει στις 29 ε, Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν οι συντονιστές των δύο αυτών επιτροπών αποφάσισαν να λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση την Πέμπτη από τις 8-9 το πρωί και θα σας ε, διανύμουμε σύντομα την ημερήσια διάταξη. Αυτά είχα να σας πω τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Τώρα είμαστε στο σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη, αν μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη 26η και 27η Σεπτεμβρίου, 10 και 11 Οκτωβρίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7 τη σημερινή διάταξη που είναι τα περίφημα PRIPS. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει προτείνει να αλλάξει η ημερομηνία εφαρμογής στο σχετικό κανονισμό μετά την ε, αντίρρηση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβρη. Το Συμβούλιο ήδη σε επίπεδο Κορεπέρ έχει πει ότι δεν προτίθεται να τροποποιήσει την πρόταση της Κομισιόν ούτε να την απορρίψει. Στο δικό μας το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου καλέσαμε την Κομισιόν να αναβάλει την ημερομηνία εφαρμογή των ΠΡΙΠΣ χωρίς άλλες αλλαγές στο επίπεδο υπαριθμών 1. Άρα δηλαδή θα προχωρήσουμε με βάση τον κανονισμό 51 που σημαίνει ότι τώρα η συγγήτρια θα μας παρουσιάσει τη δική της την πρόταση και θα ακούσουμε για λίγο και την άποψη των σκιωδών και των πολιτικών ομάδων ε, και μετά από αυτή τη συζήτηση ίσως ε, μπορούμε να εγκρίνουμε το κείμενο χωρίς περαιτέρω τροποποίηση. Αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην κυρία Περέσου ε, την εισηγήτρια. Κύριε σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η εξέταση θα είναι σύντομη. Αφού σχεδόν με καλύψατε, ε, είπατε όλα όσα θα έπρεπε να πω εγώ για τη διαδικασία αυτή. Έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα στις 14 Σεπτεμβρίου και θέλω να υπενθυμίσω την παράγραφο 4, διότι είναι η επιμαχή παράγραφος, στην οποία αναφερόμαστε και στις αιτιολογικές μας αναφορές. Λέγει λοιπόν ρητός η παράγραφος 4 ότι δεν επιθυμούμε να ξανανοίξουμε την νομοθεσία του πρώτου επίπεδου. Εκτός ε, εάν ε, πρόκειται μόνο για την αναβολή της ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του κανονισμού. Διότι αυτό τον καιρό και έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν έχουμε αρτίες. Ελπίζουμε το κείμενο αυτό να μπορέσει να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες, όπως μάλλον συνέβη και στο Κορεπέρ και θα μας τα επιβεβαίωσει το Συμβούλιο. Στη μήνυ σύνοδό μας τώρα την ερχόμενη 5η, του μηνός Δεκεμβρίου, έτσι ώστε το συντομότερο να λάβουμε τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ αυτό το ενημερωτικό ε, κείμενο που είναι τόσο σημαντικό για τους ε, ιανικούς επενδυτές, τους μικροεπενδυτές επίσης λεγόμενους. Βλέπω τον κύριο Μπάλτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι ακόμα πιο σύντομος από τη συνάδελφο Μπερές. Ε, και εμείς υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να εγκριθεί όλο αυτό με τη μορφή που το προτείνετε εσείς. Το υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να δούμε και να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γρήγορα να καταθέσει προτάσεις της. Ευχαριστώ. Η ΣΥΑΡ, κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ τι να προσθέσω. Δεν έχω πολλά να πω. Με κάλυψαν οι συνάδελφοι, συμφωνώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε. Για την κατεξοδότηση πράξη για τις εξουσίες ε, παρέμβασης που δημοσιεύθηκε στις 29 Οκτωβρίου κάτι στην ε, επίσημη εφημερίδα. Και παρόλο που θα τεθεί σε ισχύ αργότερα ο κανονισμός πρίπς μετά την περαιτέρω συμπληρωματική ε, κατεξουδότηση πράξη για τις ε, ε, εξουσίες επέμβασης. Αυτό θα προκαλέσει νομική ανασφάλεια για τους ε, κατασκευαστές κατά τη διάρκεια της περίοδου παρέμβασης και πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους καθησυχάσει σε σχέση με τις δυνατότητες και εξουσίες αυτές. Δηλαδή από τις 31 Δεκεμβρίου φέτος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βγάλει οδηγίες για τις εθνικές εποπτικές αρχές, ποια θα είναι η διαδικασία, ρωτώ. Ευχαριστώ. Yeah. Thank you, of course. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτή η πρόταση που συζητάμε απλά εξετάζει τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού. Δεν ξέρω. Η Επιτροπή θέλει να λάβετε το λόγο. Παρακαλώ. Για να απαντήσετε στην ερώτηση. Δεν βλέπω κανείς άλλος. Θέλετε κι εσείς να λάβετε το λόγο, κύριε Λάμπερτς. Σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έβλεπα τι συνεδρίες από τον διάδρομο και νόμιζα ότι θα τη γλιτώσω αλλά τέλος πάντων επειδή είδα ότι ε, μείνατε εδώ κάποιοι στάντηκα ε, το αίσθημα καθήκοντας με οδήγησε στο να έρθω εδώ γιατί νομίζω ότι και ο Σβέν θα ερχόταν αν είχε μείνει εδώ πρώτον στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για μια ταχεία ε, ρύθμιση αλλά στο βαθμό που περιορίζεται στη αναβολή κατένα μόνο έτος όπως γνωρίζετε έχουμε συμφωνήσει με το ψήφισμα ψήφισμα που λέει να απορριφθεί το αρχικό σχέδιο και το κείμενο του επίπεδου 1 να παραμείνει ω έχει. Η δυνατότητα αυτή της ταχείας ρύθμισης είναι μια δυνατότητα για να αλλάξει το αρχικό κείμενο. Τέλος, ο λόγος γιατί απέριψα και το σύστημα αυτό είναι ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προτινόμενων λύσεων κάτω από το πρίσμα της προστασίας του καταναλωτή. Νομίζουμε ότι η Κομισιόν έχει προτείνει ε, εξετάσεις ε, ε, που έχει προτείνει αλλαγές που είναι σημαντικές και αυτός ο ένας επιπρόσθετος χρόνος θα επιτρέψει να εφαρμοστεί καλύτερα η προτινόμενη οδηγία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εμείς ευχαριστούμε που δεν πήγατε στο πάρτι απ' έξω και που ήρθατε στη δική μας τη συνεδρίαση. Η Επιτροπή παρακαλώ έχει το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το θέμα της, ε, των ε, αρμοδιοτήτων εφαρμογής. μπήκε για πρακτικούς λόγους. Έχουμε μελετήσει το τι γίνεται με την ημερομηνία για την θέση ισχύ. Δεν, ε, α, δεν προτείναμε, προτείναμε την αλλαγή για το επίπεδο 1. Οι νομικοί μας είπαν ότι για το επίπεδο 2 δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Οπότε έπρεπε να, πρέπει να καθυστερήσει και για το επίπεδο 2 η θέση σε εφαρμογή όπως γίνεται για το επίπεδο 1. Και επίσης, στα όσα είπε ο κ. Λάμπερτς, δουλεύουμε πολύ στενά για τα τέσσερα σημεία βεβαίως που αναφέρονται στο ψήφισμα για τα διάφορα σενάρια που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε υπό το φως αυτής της συζήτησης νομίζω ότι μπορώ να σας προτείνω σύμφωνα με το άρθρο 50 1 να εγκρίνουμε το κείμενο χωρίς τροπολογίες. Το άρθρο λέει, μετά την πρώτη συζήτηση, ε, ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει αν, ε, να υπάρξει υιοθέτηση εκτός, χωρίς τροπολογίες εάν τα μέλη της Επιτροπής έχουν ε, αντίρρηση. Ο πρόεδρος θα υποβάλει την πρόταση αυτή σύμφωνα με τον κανόνα 150, σημείο 1, δεύτερη παράγραφος. Οπότε, δεν βλέπω να έχουν τα μέλη κάποια αντίρρηση. Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κείμενο εγκρίνεται χωρίς τροπολογίες και θα υποβληθεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν την ε, συζήτηση. Αύριο το πρωί θα ξαναξεκινήσουμε στις 9. Πέρασε συνεδρίαση.